Yeah. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε υποψήφιε επίτροπε, κύριε Μποητικόφσκι, κυρίες μου και κύριοι, σας ε, καλωσορίζω, αγαπητέ κύριε Βοητσεκόφσκι, εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής ε, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπωσδήποτε η παρουσία σας είναι μια σημαντική στιγμή για την Επιτροπή μας και βεβαίως ε, ε, βρίσκεστε και σε γνωστά λιμέρια. Ήσασταν μέλος αυτής της Επιτροπής για 12 χρόνια και ήσασταν ε, και αντιπρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής αυτής πριν εγκαταλείψετε το Κοινοβούλιο για να γίνετε τα τελευταία τρία χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν επικεντρωθείτε στα ευρωπαϊκά είχατε μια καριέρα δικαστικού στην χώρα σας μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως παίξετε σημαντικό ρόλο ως ε, βουλευτής ε, γενικός ε, γραμματέας στην Πολωνία για ζητήματα νομοθετικά και δικαστικά και θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως το Κοινοβούλιο με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν για τη εξαγωγή των ακροάσεων θα σας κρίνει με βάση των ικανοτήτων σας, της προσήλωσής σας στην ευρωπαϊκή ιδέα και την ε, ανεξαρτησία σας ε, βεβαίως ε, και βεβαίως την γνώση του χαρτοφυλακίου και τη δυνατότητα επικοινωνίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ο κύριος Βοητεκόφσκι έχει απαντήσει γραπτός ε, στο ερωτηματολόγιο. Οι γραπτές απαντήσεις έχουν ήδη μοιραστεί σε όλους τους βουλευτές, ε, σε όλες τις γλώσσες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, ο Επίτροπος, ο υποψήφιος ο Επίτροπος κ. Βοητσακόφσκι, να σας υπενθυμίσω πως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει ε, κάποια αντίρρηση για την διεξαγωγή της ακρόασης. Πριν τώρα περάσουμε στην συζήτηση, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την διεξαγωγή της συζήτησης. Ο οριστής επιτροπός ε, θα κάνει μια αρχική δήλωση που δεν θα διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Στο τέλος ε, της συνεδρίασης θα έχει 5 λεπτά χρόνο για μια δευτερολογία. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βοτσεχόφσκι για το... Θα σεβαστείτε τον χρόνο αυτό. Μετά από την εισαγωγή θα υπάρξει χρόνος για 25 ερωτήσεις των βουλευτών. Η συζήτηση αυτή θα γίνει σε 5 λεπτά και ε, σε τρία λεπτά, είναι λεπτό η απάντηση, δύο λεπτά η απάντηση του κυρίου Βοτσεχόφσκη. Η κάθε ερώτηση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από ένα λεπτό, συν ένα λεπτό η επερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και παρακαλώ τους συναδέλφους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα. Ο πρώτος γύρος 7 ερωτήσεων θα είναι από τους συντονιστές των ομάδων. Ο δεύτερος γύρος 18 ερωτήσεων είναι μοιρασμένο μεταξύ των ομάδων συν ε, ενό εκπροσώπου των μη εγγεγραμμένων βουλευτών. Σας παρακαλώ να έχετε κατά νου πως υπάρχει διερμηνία στις 23 γλώσσες, οπότε μπορούν όλοι να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Όμως, σας υπενθυμίζουμε πως πρέπει να μεταφραστούν αυτά τα οποία λέτε, οπότε σας παρακαλώ μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ja. Gut, dann Τώρα μπορούμε να περάσουμε στις εργασίες μας, ε, κύριε Ποητεκόφσκι. Έχετε τώρα την δυνατότητα να μας κάνετε μια παρουσίαση 15 λεπτών. Έχετε τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ε, με, νιώθω, μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα τη μεγάλη πρόσκληση, πρόκληση να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, ήμουν για 12 χρόνια Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξα και Αντιπρόεδρος μάλιστα αυτής της Επιτροπής και συνεργαζόμαστε στενά με πολλούς από εσάς τουλάχιστον. Τα τελευταία τρία χρόνια τα πέρασα στο ελεκτικό συνέδριο και μάλιστα με τομέα αρμοδιοτήτων στο ελεκτικό συνέδριο τη Γεωργία. Και πέρυσι παρουσίασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εκθέσεις ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου για το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες και την ε, αγροτική ανάπτυξη. Επίσης, ε, έχω υποβάλει εκθέσεις για την επιστηστική ασφάλεια και τότε την έκθεση αυτή, παρόλο που την είχα ετοιμάσει εγώ, που ήταν η διασυνοριακή ε, παροχή υγειονομικής περίθαλψη, έγινε η παρουσίαση από άλλο συνάδελφο, γιατί εγώ τότε είχα ε, ε, διοριστεί υποψήφιο ε, επίτροπο. Αλλά στο μεταξύ είχα κάνει και άλλη έκθεση για τη μικροβιακή εντοχή που θα υποβληθεί στην ε, Επιτροπή Γεωργία. Όπω σα είπα, είχα, σας είχα παρουσιάσει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το πρόγραμμα για του νεαρού Αγρότε. και τότε είχα παρουσιάσει κάποιε οκαριστικέ για κάποιου τουλάχιστον πληροφορίε. Είπα ότι για μία δεκαετία, αυτό ήταν το πόρισμα της έκθεσης, ότι από το 2005 μέχρι το 2015 χάσαμε περίπου 4 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν 15 περίπου εκατομμύριο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και μετά από μία δεκαετία ήταν λιγότερο από 11 εκατομμύρια οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του τέστην. 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσει, να χάνουμε τη δεκαετία, σημαίνει ότι χάνουμε 400.000 ε, εκμεταλλεύσει το χρόνο, πάνω από 30.000 εκμεταλλεύσεις ε, το μήνα και πάνω από 1.000 ε, αγροτικέ εκμεταλλεύσει χάνονται τη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή μα συζήτηση θα κρατήσει τρει ώρε που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια τη δημόσια ακρόσης πάνω από 100 αγρότες θα χάσουν τη δουλειά τους, θα χάσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση, κάτι που θα έχει τραγικές συνέπειες στη ζωή τους. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κανείς σήμερα αγρότης και αύριο να χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Να, να γίνει ταξιτζής για παράδειγμα. Για πολλούς αγρότες είναι τραγική η κατάσταση που βιώνουν και η απειλή της απώλειας της εκμεταλλευσής τους. Γνωρίζουμε ότι στη Γαλλία είναι οξύ το πρόβλημα των αυτοκτονιών γεωργών. Και μάλιστα έγινε και μια ταινία με βάση μια αληθινή ιστορία ο άνθρωπος της γης, μια τραγική ιστορία ε, μιας γαλλικής οικογένειας που έχασε το εισόδημά της, έχασε την αγροτική της εκμετάλλευση, έχασε τη δουλειά της και μπορεί να σας ακούγονται απεσιόδοξα αυτά που λέω στην αρχή της προφορικής μου δήλωση, αλλά σας υπόσχομαι ότι ω επίτροπο Γεωργίας θα είμαι πιο αισιόδοξο. Βέβαια, ποια είναι η διαφορά μεταξύ απεσιόδοξου και αισιόδοξου. Λένε ότι ο απεσιόδοξο είναι καλύτερα ενημερωμένο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είναι κανείς ενημερωμένο να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση και να έχει μια σωστή εικόνα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας σήμερα. Και ένας από τους λόγους που αποδέχθηκα την υποψηφιότητα για το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποδέχθηκα την πρόταση που μου έγινε να είμαι υποψήφιος Επίτροπος Γεωργίας είναι γιατί βλέπω την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και αυτό θα είναι ε, ένα από τα καθήκοντα που μου ανέθεσε η εκλεγμένη πρόεδρος Φοντερ Λάιεν όπως φαίνεται και στην επιστολή των αρμοδιοτήτων που έστειλε. Οπότε, αν με εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα από τα καθήκοντά μου θα είναι να διαμορφώσω μια μακροπρόθεσμη προοπτική και όραμα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γιατί έχουμε τέτοιε μακροπρόθεσμε προοπτικέ για την κλιματική πολιτική, για την ενεργειακή πολιτική, αλλά μακροπρόθεσμη προοπτική, μακροπρόθεσμο όραμα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν έχουμε. Και είναι σημαντικό να έχουμε ένα τέτοιο μελλοντικό όραμα, γιατί οι αγρότε μα ρωτάνε Ποιο θα είναι το μέλλον μας, ποιο θα είναι ε, το μέλλον των παιδιών μας. Και είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό και να τους απαντήσουμε καταφατικά, να τους πούμε ότι ναι, υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και για να διαμορφώσουμε ένα μακροπρόθεσμο, μακρόπρονο όραμα για τη Γεωργία είναι σημαντικό. Και να προσθέσω και μία παρατήρηση. Τέτοιο όραμα είχαν ε, ηγέτες όπως ο πρόεδρος Δεκόλ, ο Κόνεραντ Αντανάουερ, ο πρωθυπουργός Αρχάνη που ήταν ε, ηγέτες όταν ε, ξεκίνησε το 1962 η κοινή γεωρική πολιτική που είναι μια επιτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στην κοινή γεωρική πολιτική έχουμε γεωργία, έχουμε επισητιστική ασφάλεια γενικώ εξασφαλισμένη ασφάλεια των τροφίμων. Βέβαια υπάρχουν και αδυναμίες. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πάντως γενικώ ήταν επιτυχημένη η κοινή γεωργική πολιτική και το 62 όταν διαμορφώθηκε το όραμα αυτής της κοινή γεωργικής πολιτικής ήταν ένα μακρόπνο όραμα των ε, πολιτικών ηγετών που αποφάσισαν να χαράξουν μια τέτοια πολιτική. Τώρα θέλουμε ένα μακροπρόθεσμο, μακρόπνο, μακρόπνο όραμα για την πολιτική για να τη μεταρρυθμίσουμε και να εξασφαλίσουμε το μέλλον όχι μόνο των αγροτών, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι μόνο πρόβλημα των Ευρωπαίων Γεωργών και κτηνοτρόφων, είναι και πρόβλημα για την κοινωνία. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους αγρότες μας. Θα πρέπει να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία και για την κοινωνία ε, είναι θέμα επιστηστικής ασφάλειας, ε, ασφάλειας του ανεφοδιασμού σε τρόφιμα. Για την κοινωνία η γεωργία είναι πολύ σημαντική, αλλά και για τον πλανήτη η γεωργία είναι σημαντική. Η γεωργία είναι πολύ σημαντικός κλάδος για την προστασία του κλίματος, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία της βιοπικιλότητας, αλλά και για την καλή μεταχείριση των ζώων. Και αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερο, γιατί ως Ευρωβουλευτής ήμουν πρόεδρος της διακοινοβουλευτικής ομάδας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Για να διαμορφώσουμε όμως ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη γεωργία, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία σαφή εικόνα και εμπεριστατωμένη της παρούσας κατάστασης. Και από τις πρώτες δράσεις που θα αναλάβω, αν μου δώσετε την έγκρισή σας, θα είναι να εκπονήσω μια ειδική έκθεση για την παρούσα κατάσταση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Μια έκθεση που θα κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης, ε, πόσους γεωργούς έχουμε, πόσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η ηλικιακή κατάσταση των γεωργών γιατί γνωρίζουμε από την έκθεση για του νεαρού αγρότε, για το πρόγραμμα για του νεαρού αγρότε που είχα υποβάλει ω μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή Γεωργία, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ηλικιακή ανανέωση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε την κατάσταση πριν από μία δεκαετία και τώρα, για να δούμε τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ορθή και εμπεριστατωμένη εικόνα της παρούσας κατάστασης. Και αυτό θα μπορούσε να είναι καλή βάση για τον προγραμματισμό και των μελλοντικών εξελίξεων της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι έχουμε το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Green Deal, για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο. Και είμαι πεπισμένος ότι η πράσινη γεωργία, η φιλοπεριβαλλοντική γεωργία θα είναι η καλύτερη λύση για το μέλλον της γεωργίας. Μία φάρμα, μια αγροτική εκμετάλλευση που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό θα εξασφαλίσει το μέλλον της γεωργίας και τη βιωσιμότητά της. Οπότε θα προτείνουμε στήριξη στους αγρότες που προστατεύουν καλύτερα το περιβάλλον, που προστατεύουν καλύτερα το κλίμα, που βελτιώνουν τις προδιαγραφές της σωστής καλή μεταχείρισης των ζώων. Προγραμματισμός αγροτικής ανάπτυξης που απαιτεί δαπάνες τουλάχιστον 30% για το κλίμα και το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλες ευκαιρίες εδώ, κυρίως για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι αν με εγκρίνετε ως Επίτροπο θα προτείνω δράσεις που θα βοηθήσουν κυρίως τις μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους μικρομεσαίους γεωργούς και κυρίως τις οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κυρίες και κύριοι, η ιδέα μου για το μέλλον είναι να είμαι ανοιχτό στο διάλογο διάλογο μαζί σας εννοείται, διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είμαι ανοιχτό και στο διάλογο με τους αγρότες, με τις οργανώσεις γεωργών, με την κοινωνία των πολιτών, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί η πολιτική μας θα πρέπει να είναι το απάβγασμα του διαλόγου με όλους τους εταίρους μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Τη μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μακροπρόθεσμο, μακρόπνο όραμα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Να εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον για τους Ευρωπαίους αγρότες, καλύτερο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον μας και αν μου δώσετε την έγκρισή σας, θα συνεργαστώ μαζί σας και με όλους τους ενδιαφερομένους για να εφαρμόσω αυτό το μακρόπνο όραμα. Θέλω να εργαστούμε όλοι για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Vielen ε, σας ευχαριστώ κύριε Βατσεχοφσκή για την ε, παρουσίαση αυτήν. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο ομιλίας. Ε, ξέχασα κάτι πριν. Να σας ενημερώσω πως η συζήτηση αυτή μεταδίδεται ζωντανά στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε μπορείτε και να την δείτε και μετά όποτε θέλετε γιατί ταυτόχρονα εγγράφεται. Λοιπόν, ξεκινάει η συζήτηση τώρα και δίνω τον λόγο πρώτα στον κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, είπατε ότι θα ξεκινήσετε με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Για την ώρα είστε ακόμα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου και αν δω τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου πριν από ένα έτος για την ΚΑΠ και τα όσα μας είπατε μόλις τώρα εδώ πέρα και κυρίως αυτά τα οποία μας στείλατε γραπτός, ε, έχω την εντύπωση πως ε, είτε εντός ενός έτους ε, μεταβάλατε εντελώ άποψη, είτε δεν συμφωνείτε με την έκθεση την ε, περσινή, γιατί ήταν ε, πάρα πολύ επικριτική όσον αφορά τη μεταρρύθμιση. Έχετε απολύτως ε, βεβαίως δίκιο, το είπατε και στις γραπτές απαντήσεις και εδώ πέρα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τους αγρότες και βέβαια οι εξελίξεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιες επενδύσεις ε, εκτός, ε, από επενδυτές εκτός Ευρώπης που αφορούν και την αγορά γης. Ε, αυτό δεν είναι μικροκαλλιεργητές. Και βεβαίως υπάρχει και το ιστορικό μοντέλο του πρώτου πυλώνα. Λοιπόν, τι θα κάνετε για αυτά τα δύο σημεία ως Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βοτζακόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Ντόφμαν. Κοιτάξτε, έχουμε επιτάπητος ε, την πρόταση μεταρρύθμισης ε, που έχει προετοιμάσει ο συναδελφός μου, κύριος Χόγκαν. Αυτή είναι η τυπική κατάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική, εκείνη γεωργική πολιτική δηλαδή ο ε, κύριος Τσόλος ως επίτροπος ε, εφάρμοζε την πολιτική που είχε προετοιμάσει η κυρία Φίσερ Μπέλ, η προηγούμενη επίτροπος. Ο κύριος Χόγκαν ε, εφάρμοσε την πολιτική που είχε προετοιμάσει ο κύριος Τσόλος. Αν γίνω εγώ επίτροπος θα εφαρμόσω την πολιτική, την κοινή γεωργική πολιτική που θα βασίζεται στην πρόταση του κυρίου Χόγκαν. Αλλά αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε για να αλλάξουμε την πρόταση αυτή βεβαίω. Εγώ τώρα εκπροσωπώ την Κομισιόν και την πρόταση της Κομισιόν, αλλά είμαι άνοιχτος για την περαιτέρω συζήτηση για να αλλάξουμε, για να βελτιώσουμε αυτή την αρχική πρόταση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι μόνο μια αρχική πρόταση και Δεν ξέρω, ίσως να μην ήμουν σαφής στις γραπτές μου απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω τώρα σαφώς ότι ε, είμαι ανοιχτό για περαιτέρω συζήτηση για τις δικές σας προτάσεις ε, για να βελτιώσουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι η βίβλος. Μπορούμε να συζητήσουμε το πώς θα την βελτιώσουμε. και βεβαίως για το ελεγκτικό συνέδριο να συμμετείχα. Δεν ήμουν ο κύριος εισηγητής αυτής της έκθεσης, αλλά το γνωρίζω. Γνωρίζω την επικριτική... Ε, παρακαλώ συντομεύετε κύριε Ποτσοπόφσκι. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι πιο πράσινη, είπε το ελεγκτικό συνέδριο, και νομίζω θα γίνει πιο πράσινη. Η πρόταση αυτή είναι για πιο πράσινη γεωργία. Κύριε Ντόρφμαν, έχετε άλλη ερώτηση. Συγκεκριμένα για τις ιστορικές πληρωμές. Συμφωνείτε μαζί μου πως ε, το μοντέλο αυτό πρέπει να το σταματήσουμε και να βρούμε ένα άλλο μοντέλο κατανομής στον πρώτο πυλώνα. Και βεβαίως αυτό είναι ιδιαίτερος πρόβλημα στις ε, μειονεκτικές ε, περιοχές και στις ορεινές ε, περιοχές ε, οι οποίες καμιά φορά είναι πολύ ρηγμένες όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων, οπότε είναι δύο φορές μειονεκτικές. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Ντόρφμαν ότι Α, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να το βελτιώσουμε αν ε, γίνεται. Και συμφωνώ ότι υπάρχουν ε, προβλήματα των αγροτών στις ε, μειονεκτικές περιοχές όπως τις όρινες και θα πρέπει να δούμε στην Ευρωπαϊκή Γεωργία παντού. Δεν επικρατούν παντού ίδιες συνθήκες και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος ε, Πάολο Ντεκάστρο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια έκτακτη ανάγκη που εκδηλώνεται με τις ολοένα και συχνότερες κλιματικές καταστροφές που πλήττουν ε, και τους γεωργούς και όλους τους πολίτες μας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση και πολύ συντονισμένη. Αντιθέτως, η νομοθετική πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠΑ ε, που συζητιέται αυτή τη στιγμή αφήνει στα κράτη-μέλη όλες τις ευθύνες για τον προγραμματισμό μιας στρατηγικής που θα αντιμετωπίσει αυτήν την μνημειώδη ε, πρόκληση. Θα έχουμε λοιπόν εθνικά σχέδια τα οποία δεν θα βασίζονται σε ένα μενού μέτρων που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι έτσι θα αποτύχει η σημαντικότερη ευρωπαϊκή ε, πολιτική και η προστασία της υγείας ε, και των καταναλωτών ε, και του περιβάλλοντος. Αυτή η επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στο ύψος των προσδοκιών για μια Ευρώπη πιο βιώσιμη, πιο ανταγωνιστική, που θα είναι πρωταγωνίστρια στην οικολογική μετάβαση και θα συνεισφέρει σε αυτό το New Green Deal το οποίο θέλουμε. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά κύριε Βοτσεκόφσκι. Ελπίζω πως ναι. Βεβαίως οι συζητήσεις συνεχίζονται για το πόσες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πόσο, πόσες στο εθνικό. Έγινε πολλή κουβέντα και στην Επιτροπή σας, από ό,τι θυμάμαι. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, διότι διαφέρουν οι καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Διαφορετικού είδους εκμεταλλεύσεις, αγροκτήματα, σε κάποιε περιπτώσει είναι πολύ μεγάλε οι γεωργικέ εκμεταλλεύσει, σε κάποιε άλλε όλο μικρέ. Και η κατάσταση των γενεών, η ηλικία των γεωργών διαφέρει πολύ από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται και η ελαστικότητα. Επανεθνικοποίηση δεν θα την έλεγα. Έχουμε κοινούς στόχους, κοινέ παρεμβάσεις, και κοινού δείκτε. Βεβαίω ο κύριος Ντεκάστρο και όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχουν δικαίωμα στην άποψή τους και θέλω να τα συζητήσω μαζί τους. Είδαμε και τις αμφιβολίες του ελεγκτικού συνεδρίου, είδαμε ότι και εσείς έχετε κάποιους ενδιασμούς για την προσέγγιση αυτή βάση των επιδόσεων Ίσως να μην είναι αρκετό για τους ελέγχους, αλλά ένα μπορώ να σας υποσχεθώ εγώ. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η έγκριση των εθνικών στρατηγικών προγραμμάτων. Θα πρέπει η γεωργική πολιτική να είναι σίγουρα φιλικότερη προς το περιβάλλον, να λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Όμως, δεν τελειώνει εδώ η δουλειά μας περαιτέρω βελτιώσεις των προτάσεων είναι δυνατές. Συνάδελφε Ντεκάστρο, επερώτηση. Ναι, υποψήφιε επίτροπε. Δεν ε, συζητάμε την απαραίτητη ελαστικότητα για τι ε, κρατικέ παρεμβάσει στο επίπεδο τη Γεωργία. Όμω η Ευρώπη θα πρέπει να παραμένει στο πιδάλιο τη γεωργική πολιτική, όπω είπατε, με ιδιαίτερε φιλοδοξίε και επιστημονικέ. Διότι το σύστημα ελέγχου των δαπανών βάσει των επιδόσεων, αυτό που έχει υποβληθεί βάσει του delivery model που λέτε κι εσεί, το νέο μοντέλο υλοποίηση, δεν θεωρείτε ότι ε, εάν ε, βασιστούμε στο σημερινό σύστημα με συμβατότητα μόνο ως κριτήριο για το τι κάνει ο κάθε επιμέρους γεωργός, πώς θα διασφαλίσουμε την κοινή διάσταση της κοινή γεωργικής πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα έχει τον προγραμματιστικό ρόλο που της αρμόζει ε, κρατώντας τα ενία στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ε, παγκοσμίω και αντίθετα με αυτά που είπατε στι γραπτέ σα απαντήσει, μήπω χρειάζονται βελτιώσει τώρα στι ε, προσεχεί νομοθετικέ προτάσει, μήπω πρέπει οι συνομοθέτε να βρουν τώρα κάποιε λύσει για να αντιμετωπίσουμε τον αναδυόμενο κίνδυνο τη ε, επανεθνικοποίηση. Κύριε Βοτσεκόφσκι, ένα λεπτό. Είμαι ανοιχτό στο να γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό. Αλλά στην νομοθετική διαδικασία, κύριε Ντεκάστρο, ίσως να σας τα πω αργότερα, αλλά είναι υποχρέωσή μου. Είναι υποχρέωσή μου να είμαι ανοιχτό σε διάλογο μαζί σα, βάσει των αρμοδιοτήτων που μου ανέθεσε και η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ε, και με εσά πρέπει να συζητήσω και με άλλα μέλη του Κοινοβουλίου και με άλλου συνομιλητέ. Σίγουρα και η ερώτηση που θέσατε τώρα είναι ένα μέρος, είναι ένα μέρος της συζήτησης που πρόκειται να γίνει. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Μιούλα. Κύριε Βοητσεκόφσκι, στις προτάσεις σας για την, ε, και στα όσα μας υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, δεν φαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι πληρωμές προς τους γεωργούς και θα πάνε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Εσείς ως Επίτροπος πώς θα καθορίσετε την ε, μετάβαση αυτή. Είναι απαραίτητη για να καλύψουμε τις ε, ελλείψεις στην τωρινή γεωργική πολιτική. Γιατί ε, αυτοί οι κανόνες της μετάβασης είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν σωστά και βαθμίδό να περάσουν τα κράτη-μέλη στο νέο μοντέλο τη Θέλουμε να έχουμε ασφάλεια ότι η μετάβαση αυτή θα γίνει σταδιακά ε, και το νέο μοντέλο θα υλοποιηθεί σωστά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν καιρό. Κύριε Βοητσεκόφσκι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Μιούλερ. Το θέμα της κρατικής βοήθειας. Είναι θέμα του Προέδρου της Επιτροπής, της Προέδρου της Επιτροπής. Είναι κυρίως θέμα ανταγωνισμού. Και ξέρω ότι προβλήματα έχουμε με την κρατική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές παρατυπίες στον χώρο αυτό. 20% των κρατικών ελέγχων αυτών που ελέγχθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο δείξαν ότι υπήρξαν παρανομίες, πλήρω παράνομες πληρωμέ. Πρέπει να διεξάγω πόλεμο για τη γεωργία, για τη σωστή υλοποίηση των κανόνων της κοινή γεωργικής πολιτικής, της μεταρρύθμισης, θα πρέπει και είναι πολύ η δουλειά που θα γίνει για το θέμα των κρατικών επιδοτήσεων ε, στην ε, Γεωργία. Και αυτές οι προτάσεις είναι μέρος των όσων θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το συζητήσουμε στην συνέχιση τη νομοθετική διαδικασία. Η πρόταση αυτή πρέπει να ετοιμαστεί, διότι πρέπει να προβλεφθεί και συνέχεια. Η ιδέα είναι να συνεχίσουμε με την τωρινή κοινή γεωργική πολιτική, με νέο προπολογισμό όμως και νομίζω ότι την 1η Ιανουαρίου του 2022 θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Έχετε περώτηση κυρία Μίλλερ. Στις συνθήκες αναφέρεται πώς ε, οι γεωργοί διασφαλίζουν την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει το άρθρο 42 που ακριβώς υπάρχει για να τονίσει την εξαιρετική θέση των αγροτών. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς ε, θα επιτύχετε αυτούς τους στόχους με μια γενική διεύθυνση που θα έχει μείνει κούφια αν οι βασικές αρμοδιότητες πάνε στη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού πώς θα μπορέσετε να προσελκύσετε τους νέους γεωργούς και γενικά την γεωργία με τόσο νέρωμα της ε, κατάστασης. Οι δε μεταβατικοί κανόνες είναι αναγκαίοι για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα κράτη. Πηγαίνουμε από το σύστημα της ε, συμμόρφωσης στο σύστημα της απόδοσης και πρέπει να μπορέσουν να ακολουθήσουν οι διοικήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά στην προηγούμενη μου απάντηση. Αυτός ο μεταβατικός κανονισμός είναι απαραίτητος. Το χρειαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει διακοπή στην κοινή πολιτική. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί συνέχεια και η μετάβαση. Συμφωνώ πάντως απόλυτα ότι η βασική υποχρέωση και αποστολή των αγροτών με βάση τη συνθήκη είναι να εξασφαλίσουν την επιστηστική ασφάλεια, την ασφάλεια τροφίμων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και δική μας υποχρέωση, δικό μας καθήκον είναι να στηρίξουμε τους γεωργούς. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε ως πολιτικοί. Να βοηθήσουμε τους γεωργούς για να υλοποιήσουν το, το στόχο τους, την αποστολή τους. Γενικώ έχουμε επιστηστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν υπάρχει πάντα σαφήνεια. Σας ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ για ένα λεπτό. Ναι, κύριε υποψήφιε. Είπατε στις ε, απαντήσεις σας ε, πώς ε, τα πράγματα θα συνεχίσουν όλα μια χαρά και ό,τι έκανε ο κύριος Χόγκαν είναι όλα εντάξει. Αλλά συγκεκριμένα, δεν μας έχετε απαντήσει. Τι θα κάνετε για να σταματήσει η απώλεια της βιοπικιλότητας που οφείλεται στη γεωργία. Δεν δίνετε καμία απάντηση για το πώς ε, θα περιορίσετε το 40% των αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτει από τη γεωργία. Λέτε ότι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και θα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορεί να είναι απάντηση επιτρόπου αυτή, από τον οποίο αναμένω πρώτον να υποβάλει νέε προτάσεις Οπότε, συγκεκριμένα, θα το κάνετε αυτό. Μετά, ποιο είναι το δικό σας το όραμα για τη μελλοντική γεωργία. Δεν είπατε κουβέντα για τη βιολογική γεωργία. Είπατε πως πρέπει να υπάρξει μία μείωση των ζυζανιοκτών που είπε και η κυρία Φοντελάιν. Πώς θα το πετύχετε αυτό. Συγκεκριμένα πείτε μας. Ο κύριος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο να σας παρουσιάσω σε μια δίλεπτη απάντηση όλο μου το όραμα. Φυσικά κύριε Χόισλινγκ, φυσικά και θα παρουσιάσω τις προτάσεις μου και την προσέγγιση μου για τη στήριξη μιας φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας που θα σέβεται και θα προστατεύει τη βιοπικιλότητα. Για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Οι μικροκαλλιεργητές που, χρησιμοποιούσαν, ε, που χρησιμοποιούν ζωτροφές που παράγουν στην ίδια τους την ε, αγροτική εκμετάλλευση. Δεν εισάγουν ζωτροφές από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή. Αυτούς να τους στηρίξουμε. Παράγουν μόνοι τους τις ζωτροφές τους. Επίσης, θα στηρίξω, όπως σας είπα, μέτρα καλής μεταχείρισης των ζώων και αναβάθμιση των προδιαγραφών ε, για την καλή μεταχείριση των ζώων, λιγότερη πυκνότητα, να μην υπάρχει συνοστισμό των ζώων. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική μέθοδο τη ε, βοσκής στο καλοκαίρι, της βόσκησης το καλοκαίρι. Ε, ή να έχουμε χειροστρομνές για τους χείρους. Θα Υποβάλλω μέτρα για το θέμα της καλή μεταχείριση των ζώων είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Θα προτείνω φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα για μια φιλοπεριβαλλοντική γεωργία. Αυτή είναι η ιδέα μου. Αυτό είναι το όραμά μου για τη γεωργία. Σας ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ για την επερώτηση. Δεν ήταν συγκεκριμένη απάντηση, αλλά τέλος πάντων. Μιλήσατε για όλους τους αγρότες, για την ανισοκατανομή των κονδυλίων. Τι θα κάνετε για να στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο τους μικρούς αγρότες. Τι γίνεται με την εξωτερική σύγκληση. Υπάρχουν μεγάλες ε, πληρωμές ε, σε κάποιες χώρες, ενώ σε κάποιες άρες είναι κλάσμα οι πληρωμές και κατόπιν. Περικοπές στο δεύτερο πυλώνα που θα φτάσουν το 30% τι θα κάνετε. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Θα πρέπει να επενδυθούν περισσότερα στην ανάπτυξη πέθρου από ό,τι προβλέπετε μέχρι στιγμής. Κύριε Πατσεχόφσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Για να βοηθήσουμε τους α, μικροκαλλιεργητές θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα παρατηρώ ότι πολλά κονδύλια του δεύτερου πυλώνα αφορούν μια μικρή ομάδα δικαιούχων, κυρίως τους μεγαλοκτηματίες. Ένα μεγάλο τμήμα του δεύτερου πυλώνα κατευθύνεται προς ένα μικρό αριθμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τις μεγαλύτερες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο δημοκρατική διαχείριση των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα, να υποφελούνται πολύ περισσότερο, να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα. Είπα προηγουμένω. Οικολογική γεωργία, φιλοπεριβαλλοντική, βιολογική γεωργία. Αυτή είναι η κατεύθυνση και εγώ αυτή την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης θα προσπίσω. Και ο δεύτερος πυλώνας θα είναι μεγάλη ευκαιρία και για τους μικροκαλλιεργητές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νταβίτ, για ένα λεπτό. Κύριε Βοτσοχόφσκι, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής θα μεριμνήσετε ώστε οι αγρότες σε όλα τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν παρόμοιες ε, ενισχύσεις και στήριξη ανάλογα με τις συνθήκες των κρατών μελών θα σεβαστείτε τις ε, ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και τις διαφορετικές ε, συνθήκες που επικρατούν. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, θα στηρίξετε την σύναψη εμπορικών συμφωνιών που θα έχουν ως συνέπεια τη μαζική εισαγωγή γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, συμφωνία με το Μερκοσούρ, με την Ουκρανία, με το Βιετνάμ θα οδηγήσουν σε κατακλυσμό των ευρωπαϊκών αγορών με εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα. Θα στηρίξετε τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε. Δύο λεπτά, κύριε Βοτσεχόφσκι. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα του Μερκοσούρ είναι ότι και των εμπορικών συμφωνιών γενικά είπατε. Ναι, όντω, πολλοί αγρότε ανησυχούν και φοβούνται τις συνέπειες αυτών των εμπορικών συμφωνιών για ευαίσθητους τομείς ε, της γεωργίας. Μπορώ να δεσμευτώ ότι θα παρακολουθώ στενά την κατάσταση και του χρόνου, το 2020 δηλαδή, θα ετοιμάσουμε μελέτη αντικτύπου με αξιολόγηση όλων των πιθανών συνεπειών για την Ευρωπαϊκή Γεωργία της σύναψης τέτοιων εμπορικών συμφωνιών σαν, σαν τη συμφωνία με το Μερκοσούρ την εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και άλλους εταίρους. Φυσικά οι αγρότες μας δεν θα πρέπει να είναι τα θύματα των, ε, συμφωνιών, των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Και αν είναι τα θύματα θα πρέπει να τους συμπαρασταθούμε, να τους βοηθήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς της αγοράς όπως την παρέμβαση στην αγορά για να τους βοηθήσουμε. Έχουμε την εμπειρία με το ρωσικό εμπάργο. Τότε βοηθήσαμε τους αγρότες. Και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε κάθε περίπτωση εγώ θα σταθώ στο πλευρό των γεωργών, για να μην είναι οι γεωργοί τα θύματα των εμπορικών συμφωνιών. Τώρα, για τις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών, φυσικά αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, το θέμα της εξωτερικής σύγκλησης, Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, η πολιτική απόφαση που θα ληφθεί θα δείξει πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε στα θέματα της εξωτερικής σύγκλησης. Ε, αυτό το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Νταβίντ, έχετε περώτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον υποψήφιο επίτροπο αν έχει ιδέες για εναλλακτικούς μηχανισμούς, για να αποφύγουμε τον επιζήμιο αντίκτυπο των ε, εμπορικών συμφωνιών που ήδη έχουμε συνάψει. Έχετε άλλες ιδέες για την αποζημίωση των γεωργών που έχουν υποστεί ζημιές από εμπορικές συμφωνίες. Παρακαλώ κύριε Βοτσεχόφσκι. Θα πρέπει να είναι η γενική αρχή του διεθνούς εμπορίου να απαιτούνται παντού οι ίδιες προδιαγραφές. Δηλαδή να απαιτούμε από τους εισαγωγείς μας τις ίδιες προδιαγραφές που τηρούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Ήμουν αρμόδιος ε, για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και ένα από τα πορίσματα του ελέγχου που πραγματοποιήσαμε ήταν ότι κάποια εισαγόμενα προϊόντα από τη Νότια Αμερική ε, παράγονταν με τη χρήση φυτοφαρμάκων που ε, απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους μας και να χρησιμοποιούμε την αρχή της αμοιβαιότητας και να απαιτούμε από τα εισαγόμενα προϊόντα τα, τις ίδιες προδιαγραφές που επιβάλλουμε στα τοπικά ευρωπαϊκά προϊόντα. Ευχαριστώ κύριο Κούζμιουκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, την, ε, για τη δήλωσή σας. Ε, ε, μιλήσατε για τις προθέσεις για το απότερο μέλλον αλλά και για το έγκυες μέλλον. Είμαστε μεγάλη, μεγάλη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, 140 δις ε, συνολική τους αξία, αλλά αυτά για τις ε, καταργασμένες ε, μεταποιημένες ύλες. Αντίθετα, τις ακατέργαστες ύλες, οι εισαγωγές είναι 80 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές. Εκεί έχουμε πάνω από 30 δισεκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ακατέργαστων ή πρώτων υλών. Πώς θα εξασφαλίσετε την ε, επισητιστική επάρκεια των Ευρωπαίων όταν υπάρχουν τέτοια μεγάλα ελλείμματα στις εισαγωγές. Ευχαριστώ όντως. Ε, τα στοιχεία που μας δίνετε είναι ακριβή. Και η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι καθαρός εξαγωγέας ε, τροφίμων, η επιτυχία μας φυσικά στηρίζεται και στις εισαγωγές. Αυτή είναι η επιτυχία της ε, αγοραπιστιστικής βιομηχανίας βέβαια, που είναι μεγάλος εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων, αλλά το έλλειμμα ε, των πρώτων υλών και η αναγκαστική εξάρτηση από τις αγωγές είναι πρόβλημα για τη γεωργία. Πάντως, αυτό είναι απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία χρήζει μεγαλύτερης υποστήριξης, μεγαλύτερης αρρωγής για να εξασφαλιστεί η επιστηστική επάρκεια και επιστηστική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Κούσμιουκ, έχετε και περώτηση. Αναφερθήκατε στην ε, έκθεση που μας υποβάλλατε ως μέρος του Ελεκτρικού συνεδρίου. Έκθεση με θέμα το πρόγραμμα για τους νεαρούς αγρότες στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Βέβαια, η έκθεση δεν ήταν και πολύ θετική για την κοινή πολιτική. Το είπατε και στην αρχή. Είπατε ότι κάθε χρόνο ε, χάνουμε ε, εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σε 10 χρόνια χάσαμε 4 δισεκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ε, ε, οπότε ίσως τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα για να αποτρέψουμε το κλείσιμο των, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την τον εξαφανισμό των εκατομμύριων εκμεταλλεύσεων κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ρωτήσατε για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, πάρα πολύ σημαντική. Ναι, πράγματι, κατά τη διάρκεια δύο δημοσιονομικών πρόπτικων ξοδέψαμε περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τους νέους αγρότες και στο ίδιο διάστημα ο αριθμός των νέων αγροτών μειώθηκε από 3,3 εκατομμύρια στα 2,2 εκατομμύρια αγροτών ε, κάτω των 40 ετών. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία οι περισσότεροι αγρότες είναι άνω των 65, όπως στην Πορτογαλία. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία η κατάσταση είναι καλύτερη, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, και μια σχετικά καλύτερη κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να είναι ευέλικτη. Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο μέσο για το κάθε κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φλάναγκαν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές από τις ερωτήσεις που θα έκανα ήδη έγιναν, οπότε περνάω στο θέμα των εισαγωγών βοήου κρέατος, εμπορικών συμφωνιών, Μέρκοσουρ και των εκεί εμπορικών συμφωνιών, όπου τώρα έχουμε γύρω στους 300.000 τόνους βοήου κρέατος που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Υπάρχει εκεί πέρα μια ασφαλιστική δικλίδα όπως λέμε που επιτρέπεται μας επιτρέπει να επιβάλλουμε προσωρινά μέτρα εάν έχουμε αναπάντεχες αυξήσεις ε, εισαγωγών που θα βλάψουν κάποιους κλάδους. Φαντάζομαι ότι αυτό αφορά τις αναπάντεχες αυξήσεις ε, οπωσδήποτε, αλλά αφορά και μια πιθανή κρίση που θα μπορούσε να προκύψει στο τέλος ε, του μήνα, δηλαδή οι Ευρωπαίοι και μόνο στην Ιρλανδία θα χάσουν πρόσβαση σε αγορά 250.000 τόνων. Εάν δηλαδή καταλήξουμε σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία πώς θα εφαρμοστούν οι μηχανισμοί αυτοί, γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα την δική μας αγορά και μετά να δούμε τους άλλους. Ε, πώς ε, θα το κάνετε αυτό. Κύριε Βοητσεχόφσκι, έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Η απάντησή μου ίσως να μην είναι αρκετά ακριβής, αλλά μπορώ να σας πω κύριε Φλάνακαν ε, το εξή. Έχω ακούσει για τα προβλήματα των Ιρλανδών αγροτών, όχι μόνο των Ιρλανδών, όλων των παραγωγών βοήου κρέατος. Μετά τον ορισμό μου, αν με εγκρίνεται βεβαίως, θα πάω στην Ιρλανδία να δω την κατάσταση ε, αυτό προσώπως, να μιλήσω με τους αγρότες εκεί, τους Ιρλανδούς, ε, να τους ρωτήσω τι χρειάζονται το δηλώνω αυτό. Όχι μόνο τους Ιρλάνδους όμως. Θα μιλήσω λοιπόν με τους αγρότες να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ε, από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Φλάναγκαν, έχετε και άλλη ερώτηση. Ναι, ναι. Ελπίζω να το κάνετε αυτό πράγματι γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση σε σχέση με την ε, αντίσταση στα αντιμιοκρόβια τι θα κάνετε με το θέμα αυτό και θα προτείνετε κάποιες εναλλακτικές στην εντατική γεωργία. Γιατί βρισκόμαστε ακριβώς ε, στη θέση να κάνουμε κάτι. Αν δεν το κάνουμε, η ανθρωπότητα θα σας βρίζει. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας δεν θα σας ε, Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν. Κύριε Φλάναγκαν, να σας πω ότι αυτή δεν ήταν επερώτηση, ήταν μια τελείως ένα τελείως άσχετο θέμα. Κύριε Βοτσεχόφσκι βεβαίως, μπορείτε να απαντήσετε. να απαντήσω. Γιατί είναι αυτός ο έλεγχος ήταν ο τελευταίος έλεγχος για τον οποίο ήμουν υπεύθυνο και αφορούσε ακριβώς αυτό το πρόβλημα στα φάρμακα, τη μικροβιακή αντοχή στα φάρμακα και στον τομέα της γεωργίας. Δεν μπορώ να σας πω τα αποτελέσματα γιατί η επίσημη έκθεση θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα από το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό μπορώ να το πω, το γνωρίζω και πρέπει να δράσουμε για να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών στη γεωργία οπωσδήποτε. Το θέμα σας, γιατί, το ερώτημά σας τώρα για την εντατική γεωργία. Εγώ είμαι θετικός να στηρίξουμε την εκτατική γεωργία. Η εντατική γεωργία δεν είναι καλή λύση για το περιβάλλον, για το κλίμα κτλ. Ε, θα στηρίξω την εκτατική γεωργία. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος του γύρου των συντονιστών και είμαστε μια χαρά. Ακριβώς 3 και 25 όπως είχε προβλεφθεί και έχουμε φτάσει στον κύκλο των ε, επόμενων 18 ερωτήσεων και θα είμαι πολύ αυστηρός. Ε, κύριο Σόιντο, για ένα λεπτό. Το 2018 η Αμερικανική Διοίκηση επέβαλε δασμό 35% στις ε, Ισπανικές επιτραπέζες ελιές που εισήγαγε από την Ευρώπη. Ε, πλήγμα για την Ανταλουσία εκατομμυρίων ευρώ και απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Ήδη τότε είχαμε επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για μια επίθεση όχι μόνο εις βάρος της Ισπανίας, αλλά κατά του συνόλου του αγοροεπιστηστικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα ήταν η τελευταία επίθεση. Σήμερα η κυβέρνηση του Τραμπ επανέρχεται και πλήττει δεκάδες ε, τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο. Τυριά, ίνος, ελαιόλαδο, αλκοολούχα ποτά, εσπεριδοειδή. Και αν επιβεβαιωθούν οι νέοι δεσμοί, πολλέ ε, επιχειρήσει θα εγκαταλείψουν την Αμερικανική αγορά με απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασία. Η κατάσταση θα ήταν αφόρητη. Γι' αυτό λοιπόν, τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε ω επίτροπο για να προστατεύσετε τον αγροπιστιστικό κλάδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου είδου επιθέσει προστατευτισμού εκ μέρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ κύριο Βοητσεχόφσκι για δύο λεπτά. Ναι, το έχω ακούσει αυτό το πρόβλημα. Είμαι ενήμερο για το πρόβλημα αυτό και το πλήγμα που υπέστη ζήτησαν οι Ισπανοί γεωργοί. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τον Επίτροπο Χόγκαν που θα είναι αρμόδιος για το εμπόριο για να ενημερωθούμε καλύτερα για το θέμα αυτό και να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποιο μηχανισμό να βοηθήσουμε τους Ισπανούς αγρότες. Δεν ξέρω ε, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, ίσως είναι θέμα αθέμητου ανταγωνισμού, του εμπορίου. Θα δούμε, ευχαριστώ κύριε Ζωήδο που μας το επισημαίνετε, θα το συζητήσω με τον αρμόδιο επίτροπο εμπορίου. Ευχαριστώ. Υπάρχει επερώτηση κύριε Ζωήδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον υποψήφιο επίτροπο για την απάντησή του και κυρίως για την πρωτοβουλία του να συνεννοηθεί με τον υποψήφιο Χόγκαν, που μέχρι τώρα ήταν επίτροπο Γεωργία και θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου, ώστε να προλάβετε αρνητικέ εξελίξει. Πάντω, ε, δεδομένων των εξελίξεων στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία, είναι επιτακτική ανάγκη να ε, προλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναλάβει δράση πριν είναι πολύ αργά. Ένα λεπτό, κύριο Βοητσεχόφσκι. Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Ζόιδο, που μας επισημάνατε αυτό το θέμα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και θα αναζητήσουμε λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ένα λεπτό ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε υποψήφια επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να αφαιρθώ στη νέα στρατηγική που προωθεί η εκλεγμένη πρόεδρος. Η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, όπως τη λέει. Αυτά ήταν από τα θετικά σημεία που μας άφησε η κρίση των τρελών αγελάδων. Και η νέα Επιτροπή θέλει να προωθήσει με πιο ανανεωμένο και βιώσιμο τρόπο αυτή την πολιτική. Την πολιτική από το χωράφι στο πιάτο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ε, ουσιαστικής ε, επιστηστικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με την πλούσια εμπειρία που έχει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας μέσα σε επικεφαλής θα εξασφαλίσει, εξασφαλίσει συντονισμό με τι γενικέ διευθύνσει υγεία, Ανταγωνισμού και εσωτερική αγορά, Αυτό πραγματικά θα ήταν μεγάλη είδηση και για μένα και για την Επιτροπή μα. Βέβαια, στην επιστολή των αρμοδιοτήτων τα, η, γενική, η εκλεγμένη πρόεδρο ζητά από τη Γενική Διεύθυνση να συμβάλλει απλώ στη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, που σημαίνει ότι δεν θα προστατα... πρωτοστατήσετε εσείς και η Γενική Διεύθυνση άγκρι στη νέα στρατηγική. Και ποια θα είναι η τελική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πραγματικά και σημαντικό είναι και πολύ ενδιαφέρον. Η γεωργία είναι μόνο μέρος της στρατηγικής αυτής. Η υπεύθυνοι της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη ε, από την Επιτροπή θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση αυτής της στρατηγικής. Αλλά όπως είπατε, είναι στρατηγική για την ε, δημόσια υγεία, είναι και της ε, DG Sante και του ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος. Το πλέον σημαντικό ε, είναι ότι είναι σημαντικό το τι καταναλώνουμε ως τρόφιμο, τι τρώμε, αλλά και το πώς το παράγουμε, πώς παράγουμε τα τρόφιμά μας. Τι είναι η τρόπο, Η υποχρέωσή μας ως γεωργών εκτινοτρόφων και η δική μου υποχρέωση ως επιτρόπου, εφόσον με εγκρίνεται, είναι να προωθήσουμε την αιφόρο τη βιώσιμη γεωργία, ε, την παραγωγή τροφίμων που να είναι φιλική προς το περιβάλλον να επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές αλλαγές, να προάγει την υγεία των ζώων και την ευζοία. Αυτή είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους το μακροπρόθεσμο όραμά μας μας οδήγησε στις αποφάσεις, μου. Αυτός είναι ο αποφάσεις μας. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετάσχω σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Κυρία Αγγιλέρα, έχετε επερώτηση. Ναι. ναι, συμφωνούμε. Αλλά αυτό που θα θέλαμε εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας είναι ο συντονισμός αυτός για την νέα στρατηγική να αξιοποιήσει την πλούσια πείρα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας για να πρωτοστατήσετε εσείς αυτή τη στρατηγική, να μην είστε απλός ουραγός. Γιατί εδώ και χρόνια ζητούσαμε κάτι το αυτονόητο, την ε, επισητιστική πολιτική, μια πραγματική επιστηστική πολιτική. Επίσης, 10 Οκτωβρίου θα έχουμε τις διαδηλώσει ε, του Ισπανικού τομέα ελαιολάδου. Θα στηρίξετε αυτές τι πρωτοβουλίε, κύριε, Προ... κύριε υποψήφια, γιατί ο, ο προκάτοχός σας δεν τα κατάφερε. Εσείς θα εκφράσετε την υποστήριξή σα στον Ισπανικό τομέα Παραγωγή ελαιολάδου. Ευχαριστώ κύριε Βοτσεχόφσκι, ένα λεπτό. As I declared before, yes, of course, I, I can declare again. Ναι, τα, επόμενα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια έγινε σαφές οι ισπανικές προτάσεις για τους παραγωγούς είναι ενδιαφέρουσες και θέλω να εργαστώ για να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά η στρατηγική από το χωράφι στο πυρούνι του καταναλωτή, στο πιάτο, είναι σημαντική. Ε, για τη γεωργία. Το θέμα είναι κοινή διάρθρωση αυτής της πρότασης. Όμως για τη γεωργία την ίδια σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και για το περιβάλλον. Για το κλίμα. Για την βιοπικιλότητα και την προστασία της. Και στο παρελθόν κάτι κάναμε, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσιόλος για ένα λεπτό. Κύριε ε, υποψήφιε επίτροπε, συχνά διερωτώ με τι είδους συγκεκριμένο σχέδιο να χαράξουμε, να καταρτήσουμε για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους πολίτες. Τι ρόλο θα μπορούσατε να αναλάβετε εσείς εδώ, διότι οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι το θρεπτικό, τα θρεπτικά τρόφιμα, τα ποικιλία στα τρόφιμα και το να ζουν κοντά στη φύση είναι καλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε και μια αξιοπρεπή διαβίωση για τους γεωργούς. Υπάρχει ο φοβό ότι αποδυναμώνεται κοινή γεωργική πολιτική ότι οι αρμοδιότητες αρχίζουν να εκχωρούνται στα κράτη-μέλη. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε ότι πραγματικά δεσμεύεστε να εργαστείτε για να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση της ε, γεωργικής πολιτικής. Θέλουμε να ε, εργαστούμε βάσει ενός οράματος που είναι όμως και ρεαλιστικό. Και εφόσον πάρετε την έγκριση τη Επιτροπής μας για να εργαστείτε για την κοινή γεωργική πολιτική, θα συνεργαστείτε μαζί μας για να δημιουργήσετε ένα νέο όραμα για την κοινή μα πολιτική, ώστε τα τρόφιμα, παρακαλώ ολοκληρώστε, να είναι αυτά που θα θέλαμε στην παραγωγή τους. Ο κύριος Επίτροπο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Τσόλο, για την ερώτησή σας και βεβαίως και θα συνεργαστώ στενότατα μαζί σας με το Ευρωκοινοβούλιο για να έχουμε ένα μακρόπνο όραμα για τη Γεωργία. Είστε προφανώς ο πρώτος συνεργάτης που έχω υπόψη μου, εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και την υποστήριξη των πολιτών για την κοινή γεωργική πολιτική. Γενικώ υπάρχει στήριξη και κατανόηση. Περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτε καταλαβαίνουν ότι θέλουμε να, πρέπει να υποστηρίξουμε τους ε, γεωργούς μας. Είναι απαραίτητο. Όμως υπάρχει και η προσδοκία η γεωργική πολιτική να ασχολείται και με το περιβάλλον, με τις κλιματικές αλλαγές, με την προστασία της βιοποικιλότητας, ε, να μην είναι εντατική. Πολλοί φοβούνται ότι η βιομηχανική γεωργία ή εκτροφιζών είναι απειλή για το κλίμα και το περιβάλλον. Πρέπει να αποστείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα στην κοινή γνώμη. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ακολουθεί μια φιλική προς το περιβάλλον κατεύθυνση. Όσο για την επανεθικοποίηση, όπως ε, απήντησα και στον κύριο Ντεκάστρο, να συζητήσουμε και περαιτέρω διαβλέπουμε κάποιες λύσεις, αλλά κάποιες άλλες δεν έχουν σχέση με την επανεθνικοποίηση. Ε, απλώς έτσι φαίνεται. Χρειάζεται ίσως περισσότερο έλεγχο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου μαζί να δούμε πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσόλος, έχετε περώτηση. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα ακούσατε φωνέ που θα λένε ότι ή το ένα ή το άλλο δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται. Ήθελα λοιπόν μια σαφή δέσμευση από εσά. Θα δώσετε μια νέα πολιτική ορμή στην ε, κοινή αργοτική πολιτική, στην ΚΑΠ. Θα κλείσει κάποια στιγμή η συζήτηση για αυτή τη μεταρρύθμιση που συζητάμε. και θα αρχίσουμε να συζητάμε τι νέε προοπτικέ μπορούμε να δώσουμε στην ΚΑΠ. Δεν είναι μόνο το πώς θα διαιρέσουμε τον ε, ε, κουμπαρά το, το χρήμα μεταξύ των κρατών μελών. Πολλές κουβέντες έχουμε, πολλές λεπτομέρειες μας απασχολούν, αλλά εμάς μας απασχολεί το όραμα, μια θεώρηση έχετε για την πολιτική παραγωγή τροφίμων και το πώς θα πρέπει να εξοπλίσουμε τους εθνικούς πόρους. Για ένα λεπτό, κύριο Βοτσεκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω τον ενθουσιασμό να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε από κοινού ένα όραμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε το μέλλον της Γεωργίας. Ω τώρα είχαμε μόνο πενταετή πρόπτικε, διότι κάθε φορά είχαμε νέα θητεία του Κοινοβουλίου, ε, νέα θητεία τη Επιτροπή. Κάποιε φορέ φερνάγαμε και στα 7 χρόνια, όταν συζητάγαμε το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα είμαστε σε μια στιγμή κρίσιμη. Και νέο Κοινοβούλιο και νέα Επιτροπή ταυτόχρονα. Και νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και νέα γεωργική πολιτική. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε τη μακροχρόνια θεώρησή μας για την ε, Γεωργία. Σας προσκαλώ όλους να συνεργαστούμε στενά. Εάν εγκριθώ και φτάσουμε στο τέλος της θητείας μας επιτρόπου να έχουμε ένα τέτοιο όραμα, θα είναι κοινή μας επιτυχία. Σας ευχαριστούμε η κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφιο Επίτροπο. Η ε, διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών, ε, οι κλιματικέ κρίσει, το διεθνέ εμπόριο, πολλά στοιχεία που επηρεάζουν το εισόδημα των Ευρωπαίων γεωργών, συνέπειε των κλιματικών αλλαγών και τη σταδιακή ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών αγορών στι παγκόσμιε τιμέ. Οι αλλαγέ αυτέ δεν είναι χωρί κόστο. Είναι λίγοι τομεί τη γεωργία που έχουν ξεφύγει αυτό την κρίση τη πραγματικότητα που είναι σχεδόν καθημερινή σημερινή στις Βλέπουμε τι συνέπειε να καταγράφονται στι εκθέσει τη προηγούμενη θητεία τη ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Η, το πώ έχουμε θυσιάσει τι βασικέ πληρωμέ, η ενοποίηση του συστήματο Omnibus, ε, το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση σε στιγμέ κρίση, ε, σε περιπτώσει κρίση και η, η χρήση του ταμείου για τις κρίσεις τη γεωργίας. Οι ενδείξεις αυτές πάνε στην κατάλληλη, στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν είπατε τίποτα για τα θέματα αυτά ε, και μάλιστα δεν λέει τίποτα το Συμβούλιο που είναι και διχασμένο. Εσεί λοιπόν Πώ θα αναλάβετε δεσμεύσει για να εξυγχρονίσετε τα εργαλεία αυτά και να αντιμετωπίσετε το σοκ τη αγορά προστατεύοντα του γεωργού μα. Τι δέσμευση θα εκφράσετε. Κυρία Βαϊτσακόφσκι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ίσως η γραπτή μου απάντηση να μην ήταν αρκετά διαφωτιστική. Όμως μπορώ να δηλώσω, κυρία Σαντέρ, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την καλύτερη προστασία των γεωργών στην αγορά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινή αγορά. Έχουμε εμπειρία για το πώς να βοηθάμε τους ε, γεωργούς σε αυτή την περίπτωση. όπως με τις απαγορεύσεις από των εισαγωγών από τη Ρωσία και ούτω καθεξής. Θα Σαφώ θα αναλάβω δράση στον τομέα αυτό και είναι μέρο τη αποστολή μου Επιτρόπου να ενισχυθεί η αντίσταση τη δική μα τη παρουσία στι διεθνεί αγορέ. Ε, κυρία Σαντέρ, έχετε περώτηση. Θέλω να εμείνω στα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου. Τα βασικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές, τις απότομες αλλαγές, τις τιμές. Ε, τα εργαλεία αυτά εντάσσονται τώρα στο πρόγραμμα ανάπτυξη τη υπαίθρου και τα κράτη-μέλη μπορούν, αν θέλουν, να τα χρησιμοποιήσουν. Η χρήση των εργαλείων αυτών από του γεωργού δεν γίνεται συχνά γιατί κοστίζει πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ακούω αυτά που μα λέτε με προσοχή μεν, αλλά πώ συγκεκριμένα θα επενδύσετε εσεί τι προσπάθειέ σα προ αυτή την κατεύθυνση για να αναπτυχθούν αυτά τα εργαλεία σωστά. Κύριε Βοηθακόφσκι, για ένα λεπτό. Η απάντησή μου στην ερώτηση αυτή δεν μπορεί να είναι πολύ ακριβής. Ενώ ακόμη δεν έχω καν διοριστεί επίτροπος. Δεσμεύομαι όμως ότι θα συνεργαστώ με τους γεωργούς, με τα μέλη του Κοινοβουλίου, για να βρούμε καλές λύσεις. Και να ενισχύσουμε το σύστημα προστασίας των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον αναλάβω αρμοδιότητες. Αυτό μπορώ να πω τώρα ως Επίτροπος. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Αβράμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε ε, υποψήφια Επίτροπε, μας είπατε στην αρχή της προφορικής σας δήλωσης ότι Κάθε μέρα χάνουμε 4.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μέσα σε μία δεκαετία χάσαμε 4 δισεκατομμύρια και όσο διεξάγεται η ακρόασή μας, πολλοί αγρότες αντιμετωπίσουν την τραγωδία και την απώλεια της εργασίας τους. Έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ των καλών έχουμε τις κλιματικές αλλαγές, την απειλή στο περιβάλλον, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τη σχέση που έχουν οι γεωργοί με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Το αναφέρετε στις γραπτές σας απαντήσεις. Είπατε πόσο αδύναμη είναι η διαπραγματευτική θέση των γεωργών απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες διανομής και είπατε θέλετε να διορθώσετε αυτή την κατάσταση, ώστε να μην ε, είναι σε υποδέστερη θέση η γεωργία από τους ε, μεγάλους ε, από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες αλυσίδες ε, διανομής. Πώς θα διορθώσετε αυτή την ε, διαπραγματευτική αδυναμία των γεωργών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αβραμ για την ερώτηση. Πριν από 10-12 χρόνια για την ακρίβεια, το 2007, ως Ευρωβουλευτής, ήμουν από τους συντάκτες της γραπτής δήλωσης που ενέκρινε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει καλύτερα τους γεωργούς απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Και θυμάμαι ότι αυτή η πρωτοβουλία μας για να συγκεντρώσουμε υπογραφές για τη γραπτή δήλωση είχαμε λάβει την υποστήριξη πολλών οργανώσεων ε, γεωργών ε, και συνεταιρισμών γεωργικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες. Και μετά τη γραπτή δήλωση ε, ζήτησα, να ευχαριστήσω τους γεωργούς για την υποστήριξή τους και μου είπαν όχι καλύτερα κύριε Ευρωβουλευτά να μην φανεί ότι εμείς σας υποστήριξαμε γιατί φοβόταν αντίπεινα και την εκδίκηση των μεγάλων σούπερ μάρκετ, αν φαινόταν ότι ανοιχτά υποστήριζαν την γραπτή δήλωση. Και αυτή, ήταν η αυτή είναι η μακροπρόθεσμη συνέπεια των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε κανονισμό πια για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, για να αποτρέψουμε ακριβώς τέτοιες συμπεριφορές. Ως ε, αρμόδιος επίτροπος θα φροντίσω για την σωστή εφαρμογή του κανονισμού, ώστε να μην επιτρέψουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και να βελτιώσουμε τη θέση των γεωργών μας απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Κυρία Βράμ, έχετε επερώτηση? Μάλιστα. Θα ήθελα, μια και έχω την ευκαιρία, να ρωτήσω τον κύριο Βοητσεχόφσκι τι συγκεκριμένα σκοπεύει να κάνει για να βελτιώσει τη θέση των γεωργών. Και πότε θα γίνει αυτή η ευρυθής ανάλυση που είπατε για να γίνει ένας ε, απολογισμός και να έχουμε μια σαφή εικόνα τη θέση της θέσης των γεωργών απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Όπως είπα και πριν, το ζητούμενο εδώ είναι να εφαρμοστεί σωστά το νέο νομοθετικό όργανο, εργαλείο που έχουμε, που είναι ο κανονισμός για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, για την πάταξη των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και φυσικά θα πρέπει να παρακολουθούμε ε, εκ του και στην κατάσταση και σε περίπτωση που καταγγελθούν ε, αθέμητες συμπεριφορές ε, μεγάλων αλυσίδων διανομής εις βάρος γεωργών να αναλάβουμε δράση και να χρησιμοποιήσουμε τα νομικά μέσα που μας δίνει ο κανονισμός για να πατάξουμε τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν νομικά μέσα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και θα συνεργαστώ με τον αρμόδιο Επίτροπο Ανταγωνισμού και με άλλους επιτρόπους για να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αυτά προς το παρόν έχω να πω. Ευχαριστώ ο κύριος Γκερέρο. Ο κύριος Γκερέρο, κύριε Βοτσιχόφσκι, κάθεται ακριβώς πίσω σας. Κύριε Υποψήφια Επιτροπέ, δεδομένου των ανησυχιών των, ε, ανησυχιών των Ευρωπαίων για την καλή μεταχείριση των ζώων και την ε, συνεχή απειλή τη μικροβιακή εντοχή, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ξεκάθαρε πολιτικέ αλλαγέ για τον τρόπο παραγωγή των τροφίμων στην Ευρώπη, κυρίω ε, μειώνοντα δραστικά την παραγωγή, την εντατική παραγωγή θα πρέπει να μειώσουμε την εντατικότητα της ε, γεωργίας γιατί έχει ψηλά επίπεδα ρήπανσης ε, και έχουμε συστήματα που στόχο έχουν την αύξηση της ποσότητας παραγωγής αδιαφορώντας για την ποιότητα. Επίσης έχουμε μείωση του κόστου παραγωγής ε, και μη λήψη υπόψη του περιβαλλοντικού κόστους. Οπότε, σας ερωτώ, σκοπεύετε να εφαρμόσετε μια νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων. Μια και τελευταία ενημέρωση της σχετικής νομοθεσίας είναι το 2015 και πώς ε, πιστεύετε θα πρέπει να ενταχθεί ε, στην ε, νέα ΚΑΠ η καλή μεταχείριση των ζώων ενώ η Γενική Διεύθυνση Υγείας είναι η κατ' ουσίαν υπεύθυνη για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Ευχαριστώ. Για τη βελτίωση των προδιαγραφών της καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως σας είπα, αυτό το θέμα θα είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες όταν με το καλό αναλάβω. Και θα ήθελα να πω ότι έχω πείρα από τον έλεγχο ε, που έκανα ως μέλος του ελεκτικού συνεδρίου για την καλή μεταχείριση των ζώων και ήμουν ε, αρμόδιος για την πρώτη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου με θέμα την καλή μεταχείριση των ζώων. Και το πόρισμά μας ήταν ότι όταν εθαρρύνουμε τους ακτινοτρόφους να βελτιώσουν ε, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές είχαμε περισσότερα αποτελέσματα. Όχι όταν επιβάλαμε αυστηρότερα ε, πρότυπα και προδιαγραφές. Στην τρέχουσα ΚΑΠ έχουμε μέτρα καλής μεταχείρισης των ζώων. Το μέτρο υπαριθμών 14. Έχουμε και στον προγραμματισμό για την αγροτική ανάπτυξη σχετικά μέτρα. Πάντως, μέχρι στιγμής ε, τα μέτρα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. 5 δισεκατομμύρια καθ' όλη τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια για την καλή μεταχείριση των ζώων και κυρίω να ενθαρρύνουμε τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές τους. Λιγότερο εντατική κτηνοτροφία, περισσότερη βόσκηση το καλοκαίρι, χρήση χορτονομής και στις μεγάλες, στα μεγάλα χειροτροφία να χρησιμοποιούν αχυροστρομ, αχυροστρομνές για τους χείρους. Τέτοια κτηνοτροφία θέλω. Και συμφωνώ. Καλύτερα να έχουμε χίλιες φάρμες με 100 χείρους παρά μία φάρμα με 100.000 χείρους. Είναι καλύτερο και για το περιβάλλον και για το οικονομικό σκέλος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο με την δεύτερη ερώτησή του. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, βλέπουμε να υπάρχει διαρκώς όμως ε, ελλειπής ε, υλοποίηση για τα κτηνοτροφία από τα κράτη-μέλη, στα εκτροφία και βλέπουμε ότι η σύντηση, μεγάλες περιόδοι ταξιδιού, το σύστημα διοδότησης και έγκρισης δεν δίνουν τις σωστές λύσεις και η μεταφορά των ζώων των ζώων εκτό Ευρώπη πολλέ φορέ είναι ένα τρόπο να ξεπεραστούν οι ευρωπαϊκοί κανόνε. Πώ μπορούμε να χρηματοδοτούμε ακόμα τέτοιου είδου εμπόριο. Ευχαριστούμε κύριε Βοητσεκόφσκι για ένα λεπτό. Πραγματικά πολύ κύριε ερώτηση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εναλλακτικά ε, ε, συστήματα, λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Και πώς είναι οικονομικά εφικτό να πηγαίνουν ζώα από την Ιρλανδία στο ένα λιμάνι και μετά μέσα σε φορτηγό κιόλας να περνάνε με φέρι και να φτάνουν να πηγαίνουν στην, ε, στη Μέση Ανατολή. Ε, ωραία ιδέα για, την, ε, για τις εξαγωγές, αλλά εάν στηρίζουμε την κυκλική οικονομία, τους γεωργούς που παράγουν τοπικά, σε συνεργασία με τι τοπικέ βιομηχανίε. Δεν θα έπρεπε να ταξιδεύουν τα ζώα σε τέτοιε μεγάλε αποστάσει. Η παραγωγή θα έπρεπε να πηγαίνει στην τοπική αγορά. Αυτά έπρεπε να παράγουμε και τα εναλλακτικά τρόφιμα έπρεπε να υποστηρίζονται και από τι ε, ευρωπαϊκέ γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Ευχαριστούμε, κυρία Μπιτζότο. Ευχαριστώ. Όλο και πιο συχνά η γεωργία χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες ε, χώρες. Έχουμε προϊόντα όπως η ζάχαρη, το ρύζι, κρέατα, γάλας, τα, τα οποία χρησιμοποιούνται όπως είπαμε ως ε, αντάλλαγμα και επιτρέπουμε μαζικές εισαγωγές χαμηλής ε, ποιότητας που ρίχνουν τις τιμές. Σας ερωτώ λοιπόν πώς σκοπεύετε να προστατεύεστε στα επόμενα πέντε χρόνια την ανταγωνιστικότητα ειδικά των μικρών Ευρωπαίων παραγωγών και πώς σκοπεύετε να την προστατεύσετε στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες τις διάφορες ευρωπαϊκές προστατευόμενες ονομασίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε δύο λεπτά κύριε Βοητσακόφσκι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Πάρα πολύ σημαντική Πράγματι θυμάμαι ως βουλευτής ε, το ίδιο θέμα και έθεσα σε επίτροπο ε, τη δική μου ερώτηση τότε, δηλαδή το γιατί δεν προστατεύονται οι αγρότες στο διεθνές εμπόριο και η απάντηση ήταν ε, γιατί έχουμε περισσότερη βιομηχανία από τη γεωργία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αγρότες πρέπει να είναι το θύμα του διεθνούς εμπορίου. Σας δηλώνω ότι θα συνεργαστώ πολύ στενά, πρώτα απ' όλα με τον Επίτροπο, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, για να προστατεύσουμε τους αγρότες, έτσι ώστε να μην είναι το θύμα στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις άλλων συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπιζότο, Κοιτάξτε, οι διάφορες ε, διπλωματικέ διαμάχες πλήττουν συνεχώς τη γεωργία μας. Το είδαμε και με τη Ρωσία και με αλλού. Έχουμε ζημιές ε, δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για την Ιταλική ε, γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρακαλέσω να έχετε το θάρρος να υπερασπιστείτε την γεωργία εντό της Κομισιόν. Αναρωτιέμαι λοιπόν και σα ερωτώ, θα έχετε αυτό το θάρρος. και για ένα λεπτό. Η απάντησή μου θα είναι σύντομη. Ναι, θα έχω αυτό το θάρρος να προστατεύσω του αγρότε. Αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου ω επίτροπο Γεωργίας να είμαι ακριβώς ε, ο υπερασπιστής των Ευρωπαίων αγροτών όταν αυτό απαιτείται. Βεβαίω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Κυρία πολύ. Κυρία για ένα λεπτό. Και η κυρία Γκυλάρ κάθεται πίσω σας. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχω φυσικά μία ερώτηση, αλλά και τρεις ευχές. Καταρχήν θα πρέπει να έχετε ένα, ένα ανοιχτό μυαλό για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Υπάρχει μεσογειακή γεωργία, υπάρχει εντατική και εκτατική κτηνοτροφία και επίση θα πρέπει να δείξετε πυγμή ώστε να μην θυσιάσουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία μα στι εμπορικέ μα συμφωνίε. Και επίση να ταχθείτε υπέρ τη επιστήμη και τη γνώση απέναντι στην οικολογική προπαγάνδα. Και έχω μία ερώτηση που ανταποκρίνεται στην τωρινή φάση τη γεωργία. Αν έχουμε περισσότερε υποχρεώσει, περιορισμού και μικρότερου προπολογισμού, τι μέσα και νέα ενάβσματα θα δώσετε στου γεωργού για να είναι ανταγωνιστική σε όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κύριος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και των Ευρωπαίων Αγροτών θα πρέπει να τα δούμε με ανοιχτό μυαλό και σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί δεν είναι τα ίδια. Και μιλούμε μερικές φορές για την κατάσταση των γεωργών στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά οι μεσογειακοί αγρότες, οι αγρότες των από κέντρο περιοχών έχουν άλλα προβλήματα. Και θυμάμαι όταν μεταρρυθμίσαμε την αγορά ζάχαρας Πήγα στη Ρεωνιόν τότε, είχα πάει επίσης στις Κανάριες νήσους, εκεί παράγουν μπανάνες για παράδειγμα. Και υπάρχουν ε, ειδικοί τομείς στη γεωργία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τύχουν προστασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Τώρα για την οικολογία. Εγώ είμαι υπέρ της καλής μεταχείρισης των ζώων, είμαι θερμοσυπέρμαχος της καλής μεταχείρισης των ζώων και αυτό είναι από τις βασικές μου ιδέες, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν τα πρότυπα της ευζοίας και να τους στηρίξουμε στήριξη προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους για την οικειοθελή αναβάθμιση των προδιαγραφών για την ευζοία. Όχι εξτρεμιστικά οικολογικές θέσεις. Εγώ δεν είμαι εξτρεμιστής οικολόγος, αλλά η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι εκφύσεως οικολογική τομής. Άκουσα την άποψη ότι ο Γεωργός είναι ο πρώτος οικολόγος. Ο πρώτος οικολόγος ήταν Γεωργός. Θα πρέπει όμως να στηρίξουμε τους γεωργούς προς αυτή την κατεύθυνση, να τους βοηθήσουμε, όχι να τους καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Αγγιλάρ για επερώτηση. Κύριε υποψήφια επίτροπε, όπως ξέρετε, οι γεωργοί μας έχουν, χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο φυτοφάρμακα γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλά. Επίσης, έχουμε μπλοκάρει το θέμα των νέων τεχνικών βελτίωσης. Και η στοιχειώδης έρευνα για τη γεωργία γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τι ρήξη και έλευθες αλλαγές θα προτείνετε για να ανατρέψετε αυτήν την τάση. Για ένα λεπτό κύριος Βοητσεχόφσκι. Ναι, είμαι ανοιχτός και πρόθυμος για συζήτηση στο θέμα αυτό. Δεν έχω ακόμη ε, κάποια εύστοχη απάντηση στην χρήσιμη αυτή ερώτηση, θα πρέπει να το συζητήσουμε και να βρούμε καλές λύσεις. Είμαι λοιπόν ανοιχτός και διαλλακτικός και προς εσά, προς την κυρία Αγγιλέρα, προς τους ευρωβουλευτές που θέλουν συζήτηση, να την πραγματοποιήσουμε. Ευχαριστούμε κύριος Γιάννη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Στη γραπτή σας απάντηση για την μεταρρύθμιση, για τις σταδιακές ε, αλλαγέ, για το νέο σύστημα που θέλετε να δημιουργήσετε με τις απευθείας, τις άμεσες πληρωμές, ε, για να στηρίξουμε τα μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, μέχρι να αποφασίσουμε τα τρεις κοινή γεωργικής πολιτικής. Τι συμβαστικές λύσεις μπορούμε να βρούμε για τα όρια, τα ανώτατα όρια και τις ε, νέες πληρωμές για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και ποια η διαφορά μεταξύ των απευθείας πληρωμών στα κράτη-μέλη που δεν θα πρέπει να γίνονται πλέον ε, ανάλογα με τις ίσες εκτάσεις. Πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα. Ξέρουμε ότι η εντατική γεωργία είναι κάτι το διαφορετικό από και την βιομηχανική. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα με το κείμενο και τη μετάφραση. Ναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ε, εντατικής και της βιομηχανικής ε, γεωργίας. Βλέπω τι λέτε και καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα με την υπερβολικά πολύ βιομηχανική ή υπερβολικά πολύ εντατική γεωργία. Είναι παθολογικη τη γεωργία μα αυτό. Τώρα για τι διαφορέ μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη εσωτερική σύγκληση. Ε, ναι, είναι ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν στην γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για το μέλλον της ΚΑΠ. Κάποιες φορές είναι δεκαπλάσια η απόσταση ε, σε κάτω μέλο. Κάποιοι παίρνουν 100 ευρώ ένα εκτάρι και ο γείτονα 1000 για το ίδιο εκτάρι Εκτάριο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε την ε, μέτρηση και τον υπολογισμό των ποσών. Έχει να κάνει όμως με τη διαφορετική διάρθρωση των ε, αγροτεμαχίων, το διαφορετικό μέγεθος Έχουμε διαφορετική άποψη όμως και ε, είμαι ανοιχτός ε, για την κουβέντα. Πάντως με την τρέχουσα πρόταση, την πρόταση του κ. Χόγκαν, υπάρχει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετό. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω, κύριε Γιάρ. Ευχαριστούμε. Κύριε Γιάρ, έχετε ερώτηση. Με συγχωρείτε. αλλά είχα πολλά να ρωτήσω και γι' αυτό ήθελα να καταλάβω για τη σταδιακή μείωση. Έχει γίνει πολύ καιρό συζήτηση, έχουμε βρει μια συμβαστική λύση. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα, ενώ σε άλλα κάτι μέλη θέλουμε περισσότερη ευελιξία. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν εκεί. Στηρίζουμε λοιπόν τι μικρέ επιχειρήσει, λέει ένα σκέλο τη γεωργική πολιτική, αλλά αφήνουμε στου άλλου ευελιξία ώστε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο βεβαίω είναι γραφειοκρατικό πολύ, αλλά δεν, είναι, δεν θα πρέπει να είναι γραφειοκρατικό πολύ, αλλά πρέπει να προσφέρει κάποια ασφάλεια. Εσεί τι λύσει έχετε βρει για αυτή τη σταδιακή μείωση και τα ανώτατα όρια στην ΚΑΠ, τι έχετε σκεφτεί, για ένα λεπτό κύριε Βαϊτσακόφσκι. να σας απαντήσω εντάχει. Είμαι ανοιχτός για συζήτηση στο μέλλον για το σωστό συμβιβασμό. Επιτάπητος έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ ενδιαφέρουσα συμβιβαστική λύση. Ε, σε γενικές γραμμές είμαι υπέρ της ευέλικτης προσέγγισης, της ε, διαλλακτικότητας, της ευελιξίας, τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν κάπω ελεύθερα, γιατί έχουμε διαφορετικέ συνθήκε και προποθέσει. Η Δημοκρατία τη Τσεχία έχει εκμεταλλεύσει με πάνω από 130 εκτάρια μέγεθο, ενώ η Πολωνία έχει μικρά. Στην ε, Ρουμανία ακόμα μικρότερα σε εκτάρια ακόμα μικρότερε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί. Μεγάλα αγροκτήματα, μικρά αγροκτήματα. Έχουμε 80.000 αγροκτήματα με μέγεθο. Πάνω από 250 εκτάρια. 80.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνουν 22% των άμεσων πληρωμών. Των απευθεία πληρωμών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κατάινεν η οποία βρίσκεται και εκείνη πίσω από τον κύριο Βαϊτσεχόφσκι. Κύριε υποψήφια επίτροπε, ξέρουμε όλοι ότι η κερδοφόρος γεωργία και η επιστηστική ασφάλεια είναι δύο πράγματα που είναι αλληλένδετα τι θέλετε να, τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσουμε μια γεωργία η οποία να είναι κερδοφόρα και να φέρει και απαντήσει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πώ μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ μπορούμε να διαφυλάξουμε τη γεωργική παραγωγή που να είναι κερδοφόρα παντό στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ε, πιο απομακρυσμένων περιοχών αυτό που δεν είναι για δημοφιλή. Τι θα κάνετε με τι πληρωμέ για την ανάπτυξη τη πέθρου και ε, ώστε να αντιμετωπιστούν και δυσκολίε των περιοχών με γεωμορφολογικά μειονεκτήματα. Ε, το δεύτερο πυλώνα τη ΚΑΠ λοιπόν και τι άμεσε πληρωμέ. Πώ θα τον διαμορφώσετε ώστε ο οικονομικός ώστε το οικονομικό κριτήριο να μην ε, αλλοιώσει τα κριτήρια της και έρθουν να λειτουργήσουν σωρευτικά ως ε, μειονέκτημα. Κύριε Βατσακόφσκι, δύο λεπτά. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, η βιώσιμη γεωργία με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα μπορεί να είναι ανταγωνιστική εάν υποστηρίξουμε αυτό το είδος τη γεωργία. Δεν είναι θέμα να υποστηρίξουμε περισσότερο την εντατική γεωργία. Γιατί φέρνει πιο πολύ κέρδος. Μπορεί αν το βλέπει κανείς κοντόφθαλμα έτσι να είναι, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι έτσι. Και αυτό θα είναι το τίμημα εάν υποστηρίξουμε τους ε, γεωργούς που προστατεύουν το περιβάλλον μας, προστατεύουν τη βιοπικιλότητα και ούτω καθεξής. Όμως, κατά την άποψή μου, δεν την έχουμε αυτή την επιλογή. Δεν υπάρχει πια εναλλακτική. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη γεωργία που είναι φιλικά περιβαλλοντική. Και μαζί με τους γεωργούς στο πλευρό τους και όχι υποχρεώνοντάς τους να κάνουν πράγματα. Υποστηρικτικά πρέπει να λειτουργήσουμε. Αυτό είναι και το πνεύμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρώτος πυλώνας, δεύτερος πυλώνας, παντού στη γεωργική πολιτική. Ευχαριστούμε. Κυρία Κατάινεν, έχετε περώτηση. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να μιλήσουμε για, την, ε, για τα κριτήρια βιωσιμότητας και την ε, ταξινομία. Ε, εδώ πρέπει για τα κριτήρια του δεύτερου πυλώνα όμως να σκεφτούμε το εξής. Είπατε ότι οι περιοχές της Υπέθρου θέλετε να μείνουν ε, ζωντανές, ε, γεμάτες ε, δυναμισμό, όμως υπάρχει κόστος από τον δεύτερο πυλώνα. Δυστυχώς δεν έχουν όλα τα κρατημέλη τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος και θα έπρεπε να υπάρχει ίσως μεγαλύτερη ελαστικότητα στη λειτουργία μεταξύ των πυλώνων. Εσείς πώς μπορείτε να προβλέψετε αυτού του είδους την ευελιξία, την ελαστικότητα στους κανόνες κρατη μέσω του δεύτερου πυλώνα θέλουν να προβλέψουν και περιβαλλοντικά μέτρα. Κυρία Βατσεκόφσκι, ένα λεπτό για την ε, δεύτερη απάντηση. Ναι, θα σταθώ στο πλευρό των κρατών μελών που θα, κάνουν τέτοια, που θα πάρουν τέτοια απόφαση για τη μεταφορά μεταξύ πυλώνων. Και στις δι... και προς τις δύο κατευθύνσεις, από τον πρώτο ε, προς τον δεύτερο και από τον δεύτερο στον πρώτο. Είναι απαραίτητο. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες στα κάτι μελη Σε κάθε περίπτωση θα είναι εποφελές για το περιβάλλον. Και έτσι ε, θα πάει καλά η μετατόπιση κονδυλίων μεταξύ των πυλώνων. Έχετε δίκιο για το δεύτερο πυλώνα ιδίω. Στην πρόταση της Επιτροπής είχαμε περίπου 100 δις. Τώρα έχουμε λιγότερο από 80 δις. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αλλά τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα αποφασίσουν τελικά πόσο θα είναι ο, πόσο θα ο προπολογισμό στο δεύτερο πυλώνα. Φυσικά περισσότερο χρήμα σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ροντινέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, τα τελευταία πέντε χρόνια ζήσαμε έναν Επίτροπο Γεωργίας που δέχτηκε πάρα πολλές ε, κριτικές ε, γιατί τελικά αναγκάστηκε μετά από έναν πολιτικό σεισμό να διοριστεί Επίτροπος Εμπορίου. Λοιπόν, ειδικά οι αγρότες ε, οι οποίοι παράγουν ποιοτικά προϊόντα αξίζει να προστατευτούν. Στο πλαίσιο των εμπορικών ε, συμφωνιών η γεωργία ήταν το αντάλλαγμα για να αποκτήσουμε ανταλλάγματα σε άλλους ε, τομείς, χωρίς να σκεφτούμε καθόλου την κρίση που υπάρχει και την απώλεια θέσεων εργασίας. Για να υπερασπιστούμε τα μεγάλα διεθνή λόμπι, σας υπενθυμίζω πως η προηγούμενη Κομισιόν επέτρεψε την εισαγωγή ε, σιταριού με γλυφοσάτη, αδιαφορώντας για τους ε, καταναλωτές και τα τελευταία χρόνια είχαμε μια δυσανάλογη ε, αύξηση τέτοιων φαινομένων. Κύριε Βοητσεκόφσκι, παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, ε, ο δικός μου ρόλος δεν είναι να σχολιάσω το τι έκανε ο προηγούμενος Επίτροπος Η υπεράσπιση των συμφερόντων των γεωργών μας στην εμπορική πολιτική θα αποτελέσει ακριβώς αντικείμενο του νέου ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου και εκεί πέρα θα αξιολογηθεί πως έχει η κατάσταση. Αλλά μπορώ να σας πω ότι εγώ θα είμαι ένας ενεργός επίτροπος για να προστατεύσω τους γεωργούς όταν υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν θύματα διεθνών εμπορικών συμφωνιών κτλ. Θα είμαι ενεργός, οπωσδήποτε. Αυτό μπορώ να σας πω. Έχετε και άλλη ερώτηση κυρία Ροντινέλη. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Είπατε ότι θέλετε να γίνετε πρωταγωνιστής στις προσεχείς διαπραγματεύσεις, θα προστατεύσετε επιτέλους τα συμφέροντα των αγροτών. Κύριε Βοτσεκόφσκι, για ένα λεπτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Όπως είπα, το πολύ σημαντικό έγγραφο θα είναι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου. Πρώτα θα πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλες τις ε, πιθανές ε, συνέπειες που θα έχουν οι εμπορικές ε, συμφωνίες για τη γεωργία. Και μετά πρέπει να βρεθούν λύσεις μέσα για να προστατεύσουμε τους αγρότες. Γιατί βεβαίως Υπάρχουν λόγοι ε, για τους οποίους ε, γίνονται εμπορικές ε, συμφωνίες. Δεν είναι καμία τρελή ιδέα το Μερκοσούρ. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τους γεωργούς στην συμφωνία αυτή. Και έχουμε την ευκαιρία εδώ να προστατεύσουμε τους αγρότες. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε όλες τις πιθανές συνεπίσεις. Είναι πολύ σημαντική αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία θα είναι έτοιμη του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νόιχελ για ένα λεπτό. Έχω μια ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη των στόχων ε, του ΟΗΕ. Οι στόχοι 5 και 15 είναι πολύ ενδιαφέροντες. 15 στόχος προστασία των οικοσυστημάτων, προώθηση της βιωσιμότητας, καταπολέμηση της απερίμωσης, προώθηση της βιοπικιλότητας. Αυτή είναι η αποστολή μας παγκοσμίω. Εμείς με τη γεωργική πολιτική τι ρόλο παίζουμε, τι ποσοστό έχουμε σε αυτά. Να σας ρωτήσω παραδείγματος χάρη τι κάνετε για τα κριτήρια βιωσιμότητας για την εισαγωγή ζωοτροφών όπως η σόγια. Και βεβαίως υπάρχουν και τα ζητήματα τα κοινωνικά και οικολογικά. Επίσης το θέμα της αποδάσωσης, αποδάσωσης που λαμβάνει η χώρα για να φυτευτεί σόγια και άλλα προϊόντα. Οπότε οι δύο μου ερωτήσεις είναι εξή Πώς θα διασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισάγει προϊόντα που πληρούν αυτούς τους όρους και δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις και θα στηρίξετε το αίτημα του Κοινοβουλίου ειδικά για τις εισαγόμενες ε, ζωοτροφές. Κύριε Βοτσεχόφσκι, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Μιλήσατε για την εισαγωγή σόγιας. Κοιτάξτε. Είναι αναγκαίο για την κτηνοτροφία. Ε, εισάγουμε σόγια αξία 40 δισεκατομμυρίων ευρώ το έτος. Είναι μεγάλη εισαγωγές. Όπως είπα, μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες από τον δεύτερο πυλώνα, τους αγρότες που δεν χρησιμοποιούν εισαγόμενες ζωοτροφές, παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι μια πιθανή δράση και θα είναι μια πρότασή μου. Και Η βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για την γεωργία ε, και πρέπει να στηριχθεί. Αλλά συγγνώμη, ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση, γιατί την ξέχασα. Για τα δάση, για την δασοκομεία. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Και, και η απερίμωση επίσης, αυτό είπατε. Ναι. Έχουμε τη νέα έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, της προστασίας των εδαφών. Δεν υπάρχει κανονισμός ε, σχετικός. Αυτός είναι ένας λόγος για την ε, απερίμωση και η κλιματική αλλαγή βεβαίως. Οι αγρότες είναι θύματα της κλιματικής αλλαγής εν προκειμένου. Γιατί η απερίμωση είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες ε, συστάσεις και θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για την αποδάσωση. Ευτυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε... δεν έχουμε το πρόβλημα αυτό. Τα δάση τα τελευταία 20 χρόνια αυξήθηκαν κατά 11 εκατομμύρια εκτάρια. Αλλά η αποδάσωση σε άλλες υπήρους, ναι. Βεβαίω θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πρόβλημα στην διεθνή συνεργασία. Και λέει για δεύτερη ερώτηση. Παρουσιάστε την Ευρωπαϊκή Γεωργία ως θύμα. Εγώ άλλο είπα όμως. Πού είναι δράστης η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Που είναι συνυπεύθυνη για την αποδάσωση στην άλλη άκρη του κόσμου. Δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται οι εκτάσεις για να φυτέψουν σόγια πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που έχουν ε, για να καταπολεμήσουμε την κατάσταση αυτή παγκοσμίω. Κύριε Βοητσεκόφσκι για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, είναι κάπως ε, περίεργη, επίμαχη αυτή η θέση σας, ότι η γεωργία είναι υπεύθυνη, γιατί οι, οι γεωργοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ε, τα εισαγώ, τις εισαγόμενες ζωοτροφές. Αλλά και πάλι, να απαντήσω. Θα πρέπει να στηρίξουμε την κυκλική γεωργία, τοπική γεωργία. Θα είναι μια μέθοδος για να μειωθούν οι εισαγωγές από άλλες υπήρους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλινόφσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ήδη κάποιο προλαλή σα μίλησε για την εξωτερική σύγκληση, για την εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων. Τώρα, εγώ θα ρωτήσω για τι επόμενε ε, ε, δημοσιονομικές και την αιρεσιμότητα για την πρόσβαση στα κονδύλια του επόμενου ΠΔΛΤΑΠ. Ο όρος είναι η δημοσιονομική πεθερχία και το κράτος δικαίου. Αν αυτή η ρήτρα γίνει δεκτή από, τα, από κάποια κρατημέρια θα έχει τεράστιες συνέπειες για πολλούς γεωργούς που από τις άμεσες ενισχύσεις λαμβάνουν το 50% του εισοδηματός μερικές φορές. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την αιρεσιμότητα που προβλέπετε στο επόμενο ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Δεύτερη ερώτηση για τα, τα στρατηγικά σχέδια και για τη συμπερίληψη σε αυτά της έννοιας του ενεργού αγρότη που δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί μερικέ φορέ, ε, όταν κάποιο λαμβάνει μεγάλες ενισχύσει δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα γεωργό, απλώ είναι γεωκτήμονα. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πώ ορίζουν τα κράτη-μέλη τον ενεργό αγρότη. Τι γνώμη έχετε λοιπόν για αυτό το σημείο των στρατηγικών σχεδίων. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Για τον ορισμό του ενεργού αγρότη συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θέλουμε έναν γενικό ορισμό και Είμαι πρόθυμος να συνεργαστούμε στην πορεία της νομοθετικής διαδικασίας για να το συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε έναν ορισμό. Για την πρώτη σας ερώτηση, την αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου και τις δημοσιονομικές συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο, έχουμε τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό, για την πρόταση του κανονισμού δηλαδή. Και μπορώ να σας διαβάσω κάποιους τίτλους των κεφαλαίων της ε, γνωμοδότης που δεν είναι δική μου. Κάποιος συνάδελφος από το ελεκτικό συνέδριο εκπώνησε αυτή την έκθεση. Βέβαια το σύνολο του ελεκτικού συνεδρίου είναι υπεύθυνο για την έκθεση, αλλά ο συντάκτης είναι ένας. Νέες, νέοι μηχανισμοί με περισσότερη διακριτική ευχαίρεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν έγινε διαβούλευση με τους ενεχόμενους, δεν έγινε μελέτη αντικτύπου, δεν είναι σαφή τα κριτήρια και ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει σαφής υποχρέωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσει την ε, ε, πιθανότητα να υιοθετήσει μετραμετική της πρωτοβουλία. Δεν απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο των, ε, οικονομικών, των δικαιούχων και την επιρροή του εθνικού προϋπολογισμού κτλ. κτλ. Δεν είναι δικός μου ρόλος να αξιολογήσω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αλλά με βάση την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν είναι καλά ε, συγκροτημένη η πρόταση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ κύριο Καλινόφσκι για επερώτηση. Ευχαριστώ για την απόψή σας για την έννοια του ενεργού αγρότη. Ε, μάλιστα, ε, ήσταν ε, στην κυβέρνηση κατά αυτής της, αυτού του γενικευμένου ορισμού. τώρα, ε, ως Γεωργός έχω πολλές προσδοκίες ε, από σας, τον υποψήφιο επίτροπο. Και δεν θα πρέπει για τα λάθη των κυβερνώντων ε, από αμέλειες και εμένα το τίμημα να το πληρώσουν οι γεωργοί, γιατί το 50% των ε, εισοδημάτων του θα χαθεί. Και αυτό ε, επειδή το εφαρμόζουμε μόνο σε ε, μία επαγγελματική ομάδα. Αυτή είναι τεράστια πρόκληση και φροντίστε να μην γίνουν θύματα αυτής της πρότασης οι αγρότες, χάνοντας μεγάλο τμήμα των εισοδημάτων τους. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι στη νέα, συζήτηση, στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνουν ε, συζητήσεις για τη νέα πρόταση. Και επίσης ε, να εξεταστεί και η, έκθεση, η επικριτική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επικριτική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοφεύει σε αυτά τα αρνητικά σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου για την πρόταση της περιερεσιμότητας. Θα πρέπει να τα λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριος Μακάρθη, για ένα λεπτό. Commissioner, I want to refer back to your opening. Ήθελα, κύριε Πιτροπέ, να αναφερθώ στην αρχική σας δήλωση όταν είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, με το ρυθμό ε, με ρυθμό πάρα πολύ μεγάλο, εκατοντάδων χιλιάδων. Να σας εξηγήσω γιατί. Δεν είναι βιώσιμες οι εκμεταλλεύσεις, δεν βγάζουν κέρδη. Τα ήθελα λοιπόν να αναφέρω δύο τομείς ε, που πρέπει να αλλάξουν. Το πρώτο είναι η μεταρρύθμιση στις αγροτικές Σε Αυτή τη στιγμή 125.000 ε, οι πλουσιότερες ε, τέτοιες επιχειρήσεις λαμβάνουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές από την ΚΑΠ. Μιλάμε για πάνω από 10% του προπολισμού της κοινότητας ολόκληρης, όχι της ΚΑΠ. Ενώ οι περισσότεροι αγρότες λαμβάνουν ένα φιλοδόρημα. Δεύτερον, στο πλαίσιο της Γεωργίας ε, έχουμε δει μια ε, συσσωμάτωση και συγχώνευση διαφόρων αγροκτημάτων, ενώ η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα. Αυτό ρίχνει τις τιμές που λαμβάνουν οι αγρότες και έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες σε χώρες όπως η Ιρλανδία. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποια είναι τα σχέδιά σας για να υπάρξει αναδιανομή των πληρωμών και να αντιμετωπιστεί η κυριαρχία κάποιων μεγάλων εταιρικών συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη. Ε, λέγεστε Κάρθη και σας έκανα Μακάρθη. Κύριε Βοητσεκόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρθη. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ορίσει τις τιμές ε, ή την αγορά. Η αγορά είναι ελεύθερη, αλλά σε βάση περιπτώσει θα είμαι διατεθειμένος ως επίτροπος να ακούσω τους αγρότες, να δω τα προβλήματά τους και να προσπαθήσω να βρω μια λύση. Θα είμαι ο επίτροπος που θα είναι ανοιχτός για διάλογο με τους αγρότες. Αυτό σας το υπόσχομαι λέτε ότι, και έχετε δίκιο, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η διαφορά μεταξύ μικρών και μεγάλων αγροτών. Ξέρουμε ότι ένα 20% των μεγάλων εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν ένα 80% του προπολογισμού της ΚΑΠ και το υπόλοιπο 80% λαμβάνει το 20%. Πώς θα τα αλλάξουμε? Αυτό είναι ε, ένα ερώτημα που πρέπει να επιλύσουμε κατά διάρκεια της συζήτησης για το μακροπρόθεσμο όραμα για την Γεωργία. δεν υπάρχει κάποια λύση σε αυτές τις ε, πρόπτικες. Ίσως ένα πλαφόν. Ίσως ε, ενεργοί αγρότες θα μπορούσαν να είναι μια λύση. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε για το μακροπρόθεσμο όραμα της γεωργίας, δηλαδή πώς θα πρέπει να υποστηριχθούν οι εκμεταλλεύσεις, ποια είναι η θέση των μικρών εκμεταλλεύσεων, των μεγάλων. Εδώ πέρα πρέπει να βρούμε κάποιες κοινέ απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, έχετε και άλλη ερώτηση κύριε Κάρθη. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά απάντηση δεν μου δώσατε. Έχω την αίσθηση ότι ε, θα σας ε, ξαναδούμε πριν ε, τελειώσει το θέμα αυτό. Για την ώρα να σας πω δύο συγκεκριμένα πράγματα ε, στα οποία θα ήθελα την απόψή σας. Το ένα είναι το εξής. Σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό πλαφόν στις υψηλές πληρωμές για να υπάρξει μια ισορροπία για τους απλούς αγρότες. Και δεύτερον, θεωρώ πως για να αντιμετωπίσουμε την κυριαρχία ενός μικρού αριθμού ε, μέσα ζώντων πρέπει να υπάρξει απαγόρευση στην πώληση γεωργικών προϊόντων σε τιμές κάτω του κόστου. Θα στηρίξετε κάτι τέτοιο. Κύριε Βοητσακόφσκι, για ένα λεπτό. Βεβαίω ε, το dumping πρέπει να απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γενικώ. Έχω εμπειρία ως πρώην Ευρωβουλευτής ε, ότι υπήρξε μια επιτυχής ε, τέτοια δράση κατά των τιμών dumping με τις οποίες ε, εισάγονταν φράουλες από την Κίνα πριν από πολλά χρόνια, αλλά το θέμα του πλαφώνου είναι από τα πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση. Η θέση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή είναι εθελοντικό πλαφόν. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν δηλαδή. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα για το εθελοντικό ότι είναι διαφορετική η κατάσταση στο κάθε κράτος. Μεγάλες διαφορές στην κλίμακα, στο μέγεθος τον ε, αγροτημάτων. Σας είπα 30 εκτάρια είναι η μέση έκταση στη Τσεχία, 30, 10 εκτάρια στην Πολωνία. Δεν μπορεί να βρεθεί η ίδια λύση για όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι εθελοντική αυτή η πρόταση. Όχι, με συγχωρείτε, η πρόταση Κομισιόν είναι υποχρεωτική, αλλά η... αντιλαμβάνομαι την θέση που λέει ότι πρέπει να είναι και εθελοντική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καρβαλιάης τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βοτσοχόφσκι, αναγνωρίσατε εδώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές. Και μάλιστα οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι από τις περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερη προστασία και προσοχή, γιατί έχουν κάποιες διαρθρωτικούς περιορισμούς και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Βέβαια, φαίνεται ότι στο όραμά θέλετε να συμφιλιώσετε πολλές φιλοδοξίες και στόχους. Ερωτώ, ε, καλές οι φιλοδοξίες, αλλά τι συγκεκριμένα θα πράξετε για να αποκαταστήσετε κάποιες αγροτικές ζώνες που έχουν υποστεί απερίμωση, έχουν Ερημώσει, έχουν γυράσκοντα πληθυσμό, αντιμετωπίζουν και αυτές την έξοδο του πληθυσμού προς τα μεγάλα στεκά κέντρα. Οπότε, τι πρόταση θα κάνετε για τους μικροκαλλιεργητές που είναι η ραχοκοκαλιά των ε, αγροτικών ζωνών. Πώς θα τους βοηθήσετε. Ευχαριστώ κύριο Βοητσεχόφσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καρβαλιάης για την ερώτησή σας. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αγρότες αυτών των περιφερειών, των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως οι Αζόρες, η Μαδέρα, έχω πάει ε, τις έχω επισκεφτεί και άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, στην Ευρώπη, οι ισπανικές περιοχές, οι γαλλικά οι υπερπόντια διαμερίσματα, η Ρεουνιόν, η Γουαδελούπη. Είναι περιοχές, ε, η νησιά με ιδιαίτερα προβλήματα. Η πρόταση ευρωπαϊκή επιτροπή είναι να συνεχίσει την υποστήριξη, ίσως δεν αρκεί βέβαια η υποστήριξη και είμαι ανοιχτό για περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. Πάντως όταν μιλούμε για όλους τους Ευρωπαίους αγρότες, δεν ξεχνούμε τους αγρότες των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Και έχω προσωπική πείρα. Γνωρίζω μερικές από αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Μπορεί όχι όλες, αλλά τις περισσότερες έχω επισκεφτεί. Και αντιλαμβάνομαι την ιδιάζουσα κατάσταση των αγροτών τους. Ευχαριστώ κυρία Καρβαλιάης. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Μπορείτε λοιπόν να μας εγγυηθείτε ότι ε, ενστερνίζεστε τη δέσμευση του ε, Επιτρόπου Χόγκα να παρατείνετε το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ και να αποτρέψετε τις περαιτέρω περικοπές του. Μπορείτε να δώσετε στους πολίτες των εξόχων απόκεντρων περιοχών ε, αυτή την υπόσχεση ότι θα κρατήσετε και θα παρατείνετε το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ για τις περιοχές αυτές. Τα κονδύλια του ΠΟΖΕΙ έχουν υποστεί περικοπές όπως και το σύνολο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πάντως είμαι ανοιχτό και πάλι για περαιτέρω πολιτική συζήτηση και για τον γεωργικό προϋπολογισμό αλλά και για τον προϋπολογισμό του ΠΟΣΕΙ. Χρειάζεται πολιτική συμφωνία. Αν υπάρξει πολιτική υποστήριξη υπέρ τη διατήρηση των κονδυλίων του Ποζέη στα ισχύοντα επίπεδα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και καμία αντίρρηση να παραμείνει το Ποζέη αλόβητο. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Σκοτ Κάιτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βοτσεκόφσκι, ο ΙΕ έχει καταστήσει σαφέ ότι χρειαζόμαστε ω δεξαμενή άνθρακο, ω καταβόθρα άνθρακο στην ε, γεωργική μα γη. Ε, και είναι σαφέ ότι η γεωργία θα μπορούσε να μα βοηθήσει να καταπολέμησουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, αλλά όχι αν καταρρεύσει η βιοπικιλότητα. Τι εννοείται λοιπόν όταν λέτε ότι θα στηρίξετε την πράσινη γεωργία. Χρειαζόμαστε ένα βιολογικό σύστημα καλλιέργεια. Ε, εδάφη τα οποία να είναι πλούσια σε άνθρακα χωρί τη χρήση όμω φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα δάση και να πάψουμε την εισαγωγή ε, σόγια, ε, καταπολεμώντα την αποψήλωση και την, ε, την οτροφία με λάθο ζωοτροφέ. Τι θα κάνουμε λοιπόν για την προστασία τη φύση και την χρήση, την προστασία των υδάτων Πώς θα φροντίσουμε τα ψυχανθή και πώς θα, εμποδίσουμε την, πώς θα καταπολεμήσουμε τις φυσικέ καταστροφές, πώς θα είμαστε έτοιμοι να δράσουμε σε περίπτωση που προκύπτουν αυτές, πώς θα διαμορφωθεί αυτή η πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη. Ευχαριστώ, ε, κυρία Σκοτκάτο. Η απάντησή μου είναι ναι. Είμαι πλήρως έτοιμος ήταν ένας από τους λόγους Και γι' αυτό άλλωστε ήθελα και αυτή τη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πρασινίσουμε τη Γεωργία. Να πάρει μια τροπή η Γεωργία της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει πρασινότερη. Είναι πολύ σημαντικό, είναι κέριο και για τους γεωργούς είναι επίσης σημαντικό. Ακούω και αντίθετες απόψεις. Κάποιοι λένε ότι θέλω να πιθαναγκάσω τους γεωργούς στην, ε, στο πρασίνισμα της γεωργίας. Όχι, θέλω να τους ε, υποστηρίξω, να τους βοηθήσω, να σταθώ στο πλευρό τους και θέλω να βοηθήσω και όλη την κοινωνία. Ευχαριστούμε. Κυρία Σκοτκάτο, έχετε επερώτηση. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε ότι το εννοείται. Και ελπίζω να γίνει, γιατί δεν έχουμε πλέον την επιλογή να αφήσουμε τα πράγματα όπως είχαν. Ούτε για τη χρήση της γης μας, ούτε για τους γεωργούς μας. Δεν είμαστε κατά των γεωργών, είμαστε κατά των μεγάλων γεωργικών βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων που υποχρεώνουν τους γεωργούς να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες, χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν τα λοιπάσματα και μηχανές. Εμείς θέλουμε πρασίνισμα στην γεωργία, αλλά θέλουμε και έναν ε, πραγματικά ε, Εύρο στο βιολογικό τομέα στη Γεωργία με ένα πράσινο μέλλον για τη Γεωργία μα. Κύριε Βατσεκόφσκι. Συντομότερη η απάντηση. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σα. Πολύ γρήγορο. Ο κύριος Κρίστενσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα μας δώσετε τη δυνατότητα να βρούμε έναν πιο ανοιχτό τρόπο για να καθορίσουμε τι είναι μια γεωργική περιοχή ώστε να μπορεί ο κάθε γεωργός να αποφασίσει πώς θα καλλιεργεί την ε, γη του, την έκτασή του, να δώσουμε δυνατότητες καλλιέργειας της βεπικελότητας χωρίς οι γεωργοί να χάνουν ε, το εισόδημά τους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητε έχουμε για τη βιοπικιλότητα σε συνδυασμό με την πράσινη γεωργία. Πώ θα το ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί μπορούν να πετύχουν την κάλυψη τη αυξανόμενη ε, ζήτηση συγγνώμη, για τη μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνει πλούσια η παραγωγή μα, ποικίλη, και να επιτύχουμε και του στόχου του καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Είναι μέρο τη λύση η γεωργία. Κύριε Πατσακόφσκι. Ευχαριστώ Δύσκολη ερώτηση. Αλλά ποια θα είναι η προσέγγιση της γεωργίας ε, η δική μας μπορώ να πω και η δική μου προσωπικά. Τρεις σημαντικούς τομείς πρέπει να εντοπίσουμε. Όχι θέματα, τομείς. Η γεωργία και πώς θα τους στηρίξουμε, πώς θα τους προστατεύσουμε, πώς θα έχουν εισόδημα, να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στις περιοχές της Πέθρου, να είναι γεωργοί, να εξασκούν την γεωργική δραστηριότητα. Μετά για το σύνολο της κοινωνίας, επισητιστική ασφάλεια, ασφαλής τροφική αλυσίδα, Θέλουμε να είμαστε ε, διασφαλισμένοι. Είναι σημαντικότατη η πιστιστική ασφάλεια. Και το είπα και πριν. Βιοπικιλότητα, περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές. Όλα, όλα. Πρέπει να στηρίξουμε τη γεωργία. Και αυτή η υποστήριξη να είναι σε θέση να προστατεύσει όλες αυτές τις αξίες. Προστασία των γεωργών, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Αλλά να το εγγυθώ εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Για να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά την εγγύηση μόνο οι Γεωργοί οι ίδιοι μπορούν να τη δώσουν. Οι Ευρωπαίοι Γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Και να το υποστηρίξει όλη η κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κρίστανσεν, ε, επερώτηση. Ευχαριστώ. Όμως, Επίτροπε, οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφρέσουν τι θα καλλιεργήσουν στην έκτασή του, αλλά να μπορούν να καλύψουν και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. Η κυρία Φόντε Λάιεν είπε το ένας προς έναν και εγώ λέω το ένας προς δύο. Ελπίζω ότι θα είναι περιβαλλοντικά ασφαλή οι λύσει που θα βρούμε για όλα αυτά. Κύριε Βατσεκόφσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όντω, και εγώ είμαι υπέρ της, ε, του μη πολλαπλασιασμού των γραφειο, γραφειοκρατικών διατυπώσεων. Δηλαδή, όταν προστίθεται ένας κανόνα να φερούνται δύο, τι να πω. Το θέμα είναι να μην αυξηθεί η γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω με γραφειοκρατικές διατυπώσεις οι αγρότες. Αλλά έχασα το πρώτο τμήμα τη ερώτησή σα. Είχατε την καλοσύνη να την επαναλάβετε. Ε, τι, μήπως προ, προωθήσουμε μία μικρή εμβέλεια ρηπογόνα γεωργία εις βάρος της υψηλής ε, τεχνολογίας γεωργία. Εις βάρος της γεωργίας ε, υψηλής τεχνολογίας. Όχι, δεν νομίζω ότι ήμουν σαφής. Ε, με παρεξηγήσατε. Δεν είπα ότι στηρίζω μόνο τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και τις φιλοπεριβαλλοντικές επιχειρήσεις, όχι μόνο τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τις μικρές, ναι, εφόσον είναι και φιλοπεριβαλλοντικές. Θα βοηθήσουμε τους μικρούς καλλιεργητές να προετοιμαστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Το θέμα δεν είναι το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης, το θέμα είναι το είδος του τρόπου παραγωγής, το είδος της γεωργίας. Ε, ευχαριστώ. Και περνάμε στην τελευταία ερώτηση, τον κύριο Χάνσεν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού με την δέουσα επιμέλεια για τη μελλοντική ΚΑΠ πάνω από το 1 τρίτο του κοινοτικού προπολογισμού. Η ακαιρεότητά σας είχε αμφισβητηθεί το 2016 όταν οριστήκατε στο ελεγκτικό συνέδριο και πάνω από 400 ευρωβουλευτές τότε δεν σας υπερψήφισαν. Ε, διαβάσαμε προσφάτως και στο Spiegel πως είχατε κάποια προβλήματα και εκεί με τις ταξιδιωτικές δαπάνες και αναλάβω την πρωτοβουλία να επιστρέψετε 11.000 ευρώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι διπλό. Ε, συμφωνείτε ότι επιστρέψατε αυτά τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και δεύτερον Άμα δεν μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τα ταξιδιωτικά σας έξοδα, πώς θα ασχοληθείτε με το 1 τρίτο του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ, έχει τον λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο Όλαφ ολοκλήρωσε την έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016. Έλεγξαν όλες μου τις ε, ταξιδιωτικές δαπάνες, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα και επέστρεψα το ε, ποσό αυτό πέντε μήνες πριν από την έρευνα. Και η πληρωμή αυτή, ε, την οποία έκανα από μόνος μου χωρίς να μου το ζητήσουν, από το κοινοβούλιο, από την οικονομική υπηρεσία, ε, η έρευνα δεν ήταν το αποτέλεσμα, η πληρωμή δεν ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας, μάλλον ήταν η αιτία της έρευνας. Πλήρωσα με δική μου πρωτοβουλία, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να μην είναι σωστές οι πληρωμές. Ούτε ένα ευρώ κατάχρησης δεν υπήρξε. Υπάρχει και περιγραφή που έχω εδώ ε, των εγγράφων ε, του Όλαφ ε, που περιγράφουν την υπόθεση. Ε, πρόκειται για λάθη εκ που δεν επηρέασαν τον προϋπολογισμό ούτε κατά ένα ευρώ. Δεν υπήρξε καμία κατάχρηση. Το συμπέρασμα του Όλαφ επιβεβαίωσε τις δημόσιες δηλώσεις μου επ' αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Χάνσεν, με δεύτερη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είπατε επανειλημμένος, ότι το κάνατε αυθορμήτως. Δηλαδή αρνείστε ότι επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου στις 8 Ιουλίου 2014 την απόφαση του να πληρώσετε αχρεωστήτω καταβληθέντα και ότι φέρατε αντίρρηση με μια επιστολή προ του κοσμήτορε και ότι οι κοσμήτορε επιβεβαίωσαν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα το Δεκέμβριο του 2014. Γιατί όλα αυτά ήταν πριν. Δηλαδή αυτό που μα λέτε ότι το κάνατε με δική σα πρωτοβουλία είναι κάτι το διαφορετικό. Κύριε Βοητσεκόφσκι. Ε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό ήταν το θέμα του ε, περιθωρίου και έπεσα θύμα αυτής της κατάστασης. Δεν ήμουν εγώ ο δράστης. Ναι. Ήταν η πληρωμή του ταξιδιωτικού πρακτορείου και είχε... Ε, με συγχωρείτε. Θεώρησε η οικονομική υπηρεσία ότι πληρώθηκε υπερβολικά το ταξιδιωτικό πρακτορία. Αυτό δεν ήταν ε, Κάτι το οποίο έκανα εγώ λάθος. Δεν υπήρξε από μένα κάτι το μεμπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαλτσακόφσκι. Και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν στη σημερινή ακρόαση. Νομίζω πως οι απαντήσεις ε, μας βοήθησαν πάρα πολύ. και κύριε Βοητσακόφσκι, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω να κάνετε την πεντάλεπτη δήλωσή σας, αλλά πριν από αυτό να πω πως αμέσως μετά 5 και 45 με 6 και 45 θα έχουμε και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση των συντονιστών για να αξιολογήσουμε την ακρόαση. Οπότε παρακαλώ τους ε, συντονιστές να προετοιμαστούν για το εάν ο κύριος Βοητσεκόφσκι μπορεί να είναι μέλος ε, της Επιτροπής και να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Περνάμε τώρα στην πεντάλεπτη δήλωσή σας κύριε Βοητσεκόφσκι, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τις πολλές και επίκαιρες ερωτήσεις σας. Επιτρέψατε μου τώρα για να ολοκληρώσω να αναφέρω κάποια σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα ε, ε, να ε, υπενθυμίσω μια συγκεκριμένη λέξη τη λέξη διάλογος. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός στον διάλογο και θα συνεχίσω να είμαι ανοιχτός. Θα ε, είμαι σε επαφή μαζί σας, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ε, και ως άτομα και στην Επιτροπή. Και βεβαίω ο διάλογος αυτός θα επεκταθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους, με τους αγρότες, τις οργανώσεις των αγροτών και λοιπές ε, ΜΚΟ που έχουν κάποιο ενδιαφέρον στον τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε προς όφελος ε, της γεωργίας και της υπαίθρου. Δεσμεύομαι να έχουμε στις συζητήσεις σας ε, όταν το θεωρείτε αναγκαίο. Να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και θέλω να συνεργαστούμε στην ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου οράματος. Πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση για το τι χρειαζόμαστε για τους ε, γεωργούς μας ε, τις ε, δεκαετίες που έρχονται. Μια τέτοια συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο επί τη βάση μιας σωστής ανάλυσης των τάσεων και των αιτιών Ας δημιουργήσουμε λοιπόν μαζί ένα κοινό όραμα για την Ήπεθρο και την Γεωργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σύντομος. Τηρήσατε με το παραπάνω τον χρόνο. Μπορούν να χειροκροτήσουν οι συνάδελφοι. Ολοκληρώθηκε τώρα η ακρόαση. Λοιπόν, εάν οι πολιτικές ομάδες ε, το θέλουν, ε, μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα, να τα συζητήσουν σε κάποια αγωνία. Αλλά όπως σας είπα, 5 και 45 έχουμε την συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ λοιπόν τους συμμετέχοντες, τον κύριο Βόητσακόφσκι και καλό σας βράδυ.